Thank και κύριοι, καλώ ήρθατε στη συνεδρίασή μα. Θα συζητήσουμε σε λίγο την Συμφωνία σύνδεση με τη Γεωργία. Όμω σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον κύριο Κλίμκλιν, Υπουργό Εξωτερικών τη Ουκρανία σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Από το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον όσο αντιλαμβάνομαι εγώ δεν είχαμε πολύ καλά νέα. Και εγκρίνουμε από τις αντιδράσεις μετά από 3,5 ώρες συναντήσεων της κυρίας Μέρκελ, του κύριου Γιούνκερ, με την παρουσία του κύριου Πούτιν δεν νομίζω ότι μπόρεσαν να βρουν κάτι το καινούριο για να βγούμε από την κρίση. Και αν κρίνουμε και από, το, από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας χθε στη Γερμανική τηλεόραση, δεν φαίνεται να έχει προκύψει κάποιο είδους συνεννόηση η συμφωνία. και για το κατά πόσον θα πρέπει να προσφερθεί προστασία σε εκείνου που διώκονται και φωνεύονται κατά αυτόν τον φοβερό τρόπο από τις ε, πέρουσκα στραπουτεύματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Θα πρέπει να προστατευθούν οι μειονότητε. Εκφράζονται διεκδικήσεις, υποτίθεται για ιστορικές, ιστορικές διεκδικήσεις. Και πάνω σε αυτέ στηρίζονται τι στρατιωτικέ δράσει. Πάντοτε τέτοιου είδου επιχειρήματα προβάλλονταν και σε αυτά στηρίχθηκε και η, 300, η ιστορία τριών αιώνων πολέμων στην Ευρώπη. Δεν ακούσαμε δημόσια δήλωση της ε, καγκελαρίου εκτός από το ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην επεκταθεί το πρόβλημα και το κίνδυνο να πλήξει τη Γεωργία και τη Μολδαβία η κρίση. Φαίνεται να υπάρχει εδώ μια σαφή στρατηγική. Δεν ξέρω αν είστε και εσείς το ίδιο πεσιόδοξο με μένα. Αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε όταν σε μια συνεδρίαση του G20 και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνεδρίαση του G20 ε, στέλνει η Ρωσία έξι πολεμικά πλοία. στα νυχτά του Μπρίσμπεϊν. είναι προφανώς πολύ επικίνδυνη και προκλητική στάση αυτή. Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, με μεγάλη πλειοψηφία και παράλληλα με το Συμβούλιο, κυρώσαμε τη συνθήκη σύνδεσης, η συνθήκη ισχύει όσο μας αφορά πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως, όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τηρηθούν εδώ αποστάσεις και γι' αυτό σας καλώ να λάβετε το λόγο και να μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε μετά στο διάλογο μαζί σας. Παρακαλώ. Αγαπητέ Έλμερ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, πάντα, όπως και σήμερα είναι τιμή και χαρά για μένα, να μιλώ ενώπιόν σας. Έλμερ, ευχαριστώ πολύ που οργάνωσα αυτή την ευκαιρία και μου προσέφερε την ευκαιρία αυτή. Βλέπω εδώ παρόντες πολλούς από εσά που είχα την ευκαιρία να συναντήσω αμέσως μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές, πολλούς από εσά που μας υποστήριξαν. Ήσασταν παρόντες ως παρατηρητές, μας υποστηρίξατε και αυτός είναι σωστός όρος κατά τη διάρκεια των ε, της εκλογικής διαδικασίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς σαφές, το αποτέλεσμα είναι συντριπτικό. Άνω του 80% των Ουκρανών ψήφισε την, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουκρανίας, τα φιλοευρωπαϊκά κράτη. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Και σημαντικό επίσης είναι πολύ ότι δεν υπάρχει, δεν εκφράστηκε και μια πραγματική ουσιαστική διαφορά γεωγραφικά ως προς την αντίληψη των πολιτών. Οι πολίτες εκφράστηκαν με σαφή πλειοψηφία σε κάθε γεωγραφική περιοχή υπέρ της ευρωπαϊκής μας πορείας, υπέρ του ευρωπαϊκού οράματος. Και τώρα έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόσκληση, πρόκληση να προχωρήσουμε, να σχεδιάσουμε και να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, γιατί έχουμε ένα πολύ στενό αλλά και μοναδικό παράθυρο ευκαιρίας Δεν πρέπει να πει κανεί ότι επειδή η Ρωσία προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή πρέπει εμεί να σταματήσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Στον αντίον πρέπει να συνεχίσουμε. Και το σχέδιο της συμφωνίας για την κυβέρνηση συνασπισμού είναι για μένα ένα μοναδικό και φιλόδοξο έγγραφο στο οποίο καταγράφονται όλες οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει μέσα στο εγκύτατο μέλλον να υλοποιηθούν προκειμένου μέσω αυτό να υλοποιηθεί και η Συμφωνία Σύνδεσης. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς που υποστηρίξατε την διαδικασία στο σύνολό τη την ε, σειρά των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη και την κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ιδιαίτερα δε εύχομαι ότι το καλύτερο και για τους φίλους από τη Γεωργία που έχουν και εκείνη τη τιμητική του σήμερα και τις προσεχείς ημέρες. Θα έχουμε λοιπόν ένα χώρο όπου οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές μπορούν να αναπτυχθούν και να ανδρωθούν. Οι κέρυες ιδέες λοιπόν για το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις θα είναι ποιες. Θα οργανωθούν μεταρρυθμίσεις μας γύρω από τέσσερις κέρυες προτεραιότητες. Καταρχάς την καταπολέμηση της διαφθοράς της πραγματικής, την πραγματική δηλαδή καταπολέμηση της διαφθοράς, όχι μόνο μέσω της αγωγής μιας σωστής και εφρόνιμης νομοθεσίας, αλλά και με την έννοια της υλοποίησης, της εφαρμογής, της δραστηριοποίησης ε, της υπηρεσίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με την έννοια του να επιτρέψουμε στον κόσμο και στην οικονομία να λειτουργήσει με τρόπο ευρωπαϊκό. Θα έχουμε επίσης την αποκέντρωση, γιατί θα αναλάβουμε ένα νέο σύστημα ε, να προωθήσουμε, ένα σύστημα με το οποίο θα μπορούν οι πολίτες να αναλαμβάνουν και περισσότερες ελευθερίες αλλά και περισσότερες ευθύνες με... ένα σύστημα χρηστής διακυβέρνησης και ένα σύστημα που θα κριθεί από το κράτος δικαίου. Ένα σύστημα στο οποίο θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση και αναδιάρθρωση ολόκληρου του δικαιοδοτικού συστήματος και του τομέα της ε, πολιτικής ασφάλειας στην ε, Ουκρανία. Ξεκινώντας σήμερα υπογράφουμε τη συμφωνία για την ευρωπαϊκή αρρωγή στο χώρο των μεταρρυθμίσεων για την πολιτική προστασία. Θα υπάρξει μια ευρωπαϊκή αποστολή που θα μας στηρίξει θα μας προσφέρει την αρρωγή της στην αναδιάρθρωση του συστήματος. Εάν ρωτήσετε τους Ουκρανούς σε τι, ε, ε, σε τι στηρίζουν την εμπιστοσύνη τους, ε, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και το καθεξής, η απάντηση θα είναι ότι η εμπιστοσύνη έχουν στις αξίες και την εκκλησία, αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους μέσα από τους θεσμούς της κυβέρνησης, μέσα από την ε, απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών πολιτικής ασφάλειας μεταξύ άλλων και βέβαια θα γίνει στη βάση αυτών και μια σειρά οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα προγραμματιστούν και θα καταγραφούν στη μελλοντική συμφωνία για κυβέρνηση, το πρόγραμμα της κυβέρνησης, με επακριβή χρονοδιαγράμματα, όχι σχετικά από χρονοδιαγράμματα. Το δικό μου δε όραμα, το δικό μου όνειρο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει τη συνδρομή της σε κάθε τομέα των μεταρρυθμίσεων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα σε κάθε Υπουργείο. Εμπειρογνώμονες Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν σε κάθε τοπικό επίπεδο και να προσφέρουν με την υποστήριξή τους την ε, αρρωγή αυτή για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η διαδικασία αυτή για να στεφθεί με επιτυχία μπορεί να προχωρήσει εφόσον και μόνο εφόσον δεν προσπαθήσει πλέον άλλος να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας. Αυτό που βλέπουμε όμως στο Ντόνιεσκ, στο Λούγκανσκ είναι χιλιάδες ε, στρατιωτών των Ρώσων μαζί με, τους, με τις δυνάμεις των αυτονομιστών προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση. Εκατοντάδες και επαναλαμβάνω εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία περιπολούν είναι δυνατόν να αγοράσει κανείς ε, καλάσνικοφ στην αγορά και ίσως αυτό να είναι μια εύκολη υπόθεση αλλά φτάνουν και σε πολύ πιο βαρύ, βαρύ εξοπλισμό πλέον οι δυνατότητες διευκόλυνσης από την μαύρη αγορά. Έχουμε ακόμα ε, στις περιοχές του Ντούνια, Ντόνιας και του Λούγκανσκ ε, που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ακόμα τα σύνορα με τη Ρωσία περνούν ε, σε μεγάλες ποσότητες βαρέα όπλα. Και εμείς από πλευράς μας στηρούμε αμπαρεγκλήτως τη συμφωνία του Μίνσκ. Θεωρούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στην περιοχή γιατί πρέπει να αποσυρθούν οι δυνάμεις, να εξασφαλιστεί η εγγύηση, η ασφάλεια το, της διαχωριστικής γραμμής, να αποσυρθούν οι δυνάμεις, να αποφυλακιστούν, να απελευθερωθούν οι όμοιροι, γιατί έχουμε πάνω 500 ομοίρους που ζουν σε συνθήκες απάνθρωπες, που υποφέρουν, γιατί τώρα οι καιρικέ συνθήκες με τον επερχόμενο χειμώνα είναι πάρα πολύ σκληρές και οι θερμοκρασίες πολύ χαμηλές. Έχουμε όμως και πολιτικούς κρατουμένους στη Ρωσία, όπως τον Νάιτζελ Σάφτσακα, τον ήρωά μας, πιλότο αεροσκάφους και όχι μόνο αυτούς, όχι μόνο αυτούς δηλαδή που κρατούν οι Ρώσοι φυλακές τους, αλλά που έχουν απαγάγει από το έδαφος της Ουκρανίας, τους κρατούν ομήρους, τους έχουν βάλει τσουβάλι πάνω από το κεφάλι και τους έχουν μεταφέρει. Και η κατάσταση επιδεινώνεται διαρκώς σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα μετά την άσκηση στις 2 Νοεμβρίου, άσκηση που ορισμένοι στον Τόνιας και το Λούγκανσκ ε, θεωρούν ότι μπορούν να αποκαλούν εκλογική αναμέτρηση, με σαφή υποστήριξη από τη Ρωσία και την προσπάθεια να εκλεγεί ε, πρόεδρος ε, υποτίθεται και το Κοινοβούλιο για τον Τόνιας και το Λούγκανσκ, έτσι εντείνεται μία παγωμένη σύραξη, αλλά θέλω να καταλάβετε όλοι εδώ ότι το Ντόνιασκ και το Λουγκάνσκ δεν μπορούν να μετατραπούν σε μία άλλη υπερδνηστερία ή μία Απχαζία γιατί είναι τόσο δεινή η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί και επιδεινώνεται διαρκώς και γιατί είναι τέτοια η επέμβαση και η παρουσία της Ρωσίας που θα αποσταθεροποιεί τον τομέα, δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να δούμε σταθεροποίηση με όλες μας τις προσπάθειες. Αυτό λοιπόν που θα χρειαστούμε θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει με μία φωνή, να μην κατακαιρματιστεί η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις προσπάθειες της Ρωσίας και υπ' αυτή τη ενία θα είμαι ευγνώμων στον κάθε ένα και την κάθε μία από εσάς που θα μεταφέρει αυτό το πολιτικό μήνυμα και που θα διατηρήσει ε, δυνατή τη φωνή με το πολιτικό μήνυμα προς τη Ρωσία και την έκκληση να προχωρήσει στην υλοποίηση και να παραμείνει δεσμευμένη στις στη συμφωνία του Μίνσκ, στους όρους συμφωνίας του Μίνσκ, να τηρήσει την κατάπαυση πυρός, γιατί κάθε μέρα χάνουμε στρατιώτες, ανθρώπινες ζωές, λόγω των όλμων που στέλνουν, που ρίχνουν οι τρομοκράτες. Εμείς δεν, δεν αρχίσαμε ποτέ να ρίχνουμε όλμους, μόνο μία φορά ως απάντηση σε όλμους των τρομοκρατών, Εχθές δεν χάσαμε ακόμα έξι στρατιώτες και είναι χιλιάδες οι υποθέσεις, οι περιπτώσεις της παραβίασης της ανακοχής. Παραβίαση ανακοχής που γεννούν μόνο αβεβαιότητα, αλλά και αίσθηση ανασφάλειας και αβεβαιότητα στον Αντώνια και και το Λουγκάνσκ για το κατά πόσο θα μπορεί να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η ηρεμία. Αυτό που θέλουμε θα είναι ένα με μήνυμα σαφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις μας και θα επιτρέψει στην Ουκρανία να υλοποιήσει με επιτυχία τις μεταρρυθμίσεις της. Θέλουμε επίσης αποφασιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία με την έννοια της στρατιωτικής και τεχνικής υποστήριξης και δεν αναφέρομαι σε παραδόσεις ε, οπλισμού, αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό, πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό, αλλά χρειάζεται ένας πραγματικά αποτρεπτικός παράγων με τη μορφή των κυρώσεων και την ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού. Και αυτό θέλω ακριβώς να σας ε, εξηγήσω ότι δεν θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τον Τόνιας και τον Λουγκάνσκ με στρατιωτικά μέσα. Αλλά το διακύβευμα εδώ είναι ότι οι πολίτες μας υποφέρουν λόγω των επιθέσεων των τρομοκρατών. Δική μας δέσμευση αλλά και αντίληψη είναι το ότι μεριμνούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι ακόμη και με δεδομένο το ότι το Ντόνιανσκ και το Λούγκανσκ δεν μας επιστρέφουν τα οφειλόμενα για το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο και τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφήσουμε να παγώσουν με τόσο χαμηλές θερμοκρατησίες που επικρατούν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ούτε δεκάρα για το ηλεκτρικό και το φυσικό αέριο που τους ε, παραδεύουμε. Άρα, εμείς αγωνιούμε και μεριμνούμε για τους ανθρώπους αυτούς εκεί, προσπαθούμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό είναι το μέλημά μας. Να φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς που απειλούνται από τους τρομοκράτες και θα θέλαμε να ζητήσουμε οποιαδήποτε υποστήριξη μπορεί να μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και τα μέλη της μέσω αυτής της στρατιωτικής ή άλλης υποστήριξης. Ιδιαίτερα θα μεριμνήσουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και στο μέλλον και θέλουμε το δικό σας μήνυμα και τη δική σας αδιάκοπη υποστήριξη, ώστε να εξηγήσουμε και στους Ουκρανούς για κάθε κέριο σημείο ευρωπαϊκής ε, του ευρωπαϊκού μας θεματολογίου ότι αυτό ακριβώς είναι το καλύτερο. Όπως ακριβώς είναι καθήκον και δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε κάθε μία μεταρρύθμιση. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι μία ε, στήριξη αποφασιστική, απερίφραστη και μία δήλωση αφή της Ευρωπαϊκή Ένωσης για την ενίσχυση των σχέσεων και την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης, για την ε, δυνατότητα ε, ταξιδιού χωρίς υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων, για την υποστήριξη που μπορεί να μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να επισημανώ, παρακαλώ μην το θεωρήσετε απλώς συνθηματολογία, ότι εμείς αγωνιζόμαστε στην Ανατολική Ουκρανία, όχι μόνο για τον Ντόνιεσκ και τον Λούγκανσκ, όχι μόνο για την Ουκρανία. Εμείς αγωνιζόμαστε στην Ανατολική Ουκρανία για την ασφάλεια σε κάθε όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί, εάν προσπαθεί κάποιος και επιτύχει εν τέλει να δυναμητήσει την κατάσταση στο Λούγκανσκ και τον Τόνιασκ, τότε αυτό σημαίνει όχι απλώς μια μεγάλη πρόκληση, αλλά εφιάλτη για όλους μας. Για όλους μας. Πάνω απ' όλα βέβαια για την Ουκρανία, αλλά και για τον κάθε έναν και την κάθε μία από εσά. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας συντονισμένη υποστήριξη. Γι' αυτό τη θεωρούμε τόσο πολύτιμη. Υπάρχουν άλλα πολύ σημαντικά ε, στοιχεία και πορεία, η μονοπάτια που επιδιώκουμε να υλοποιήσουμε. Θέματα της οικονομίας, θέματα της ενέργειας, όπου μπορέσαμε με τριμερή μόνο εκδοχή και συνδυασμό να καταλήξουμε σε συμφωνία μόνο με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε μια πολύ σοφή απόφαση για την ενέργεια Τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε τα προβλήματα σε σχέση με την εξασφάλιση προμήθειας μέχρι το Μάρτιο σε φυσικό αέριο και να καταλήξουμε σε μια σημαντική συμφωνία για την υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης. Και θα ήθελα να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαστε ε, απαρέγκλητα προσκολλημένοι σε αυτή τη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε ούτε κόμμα ούτε τελεία. Θα εφαρμοστεί bona να καλή την πίστη, αυτή η συμφωνία και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συνολική προσέγγιση με την παροχή βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα καταφέρουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε μόνο μαζί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και με στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. I give the floor now to Mr. Plenković. Το λόγο έχει ο κύριος Πλάνκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Έλμα. Ευχαριστώ και σένα, Παύλο. τα Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ουκρανία και πρόσφατα και επίσημη ε, Επιτροπή Σύνδεσης, στην οποία θα συμμετέχω και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι βουλευτές ε, σε αυτή τη διαδικασία. Σας εγχαίρω για τον πολύ καλό και οργανωμένο τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι εκλογέ στις 26 Οκτωβρίου. διεθνώ γνωρίζετε αυτό. Αρχικά ένα ερώτημα για το πολιτικό πλαίσιο. Όλα τα βασικά ε, ε, κόμματα που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν ε, στην κυβέρνηση συνασπισμού, γιατί εμείς περιμένουμε να υπάρξει μια γρήγορη διαμόρφωση κυβέρνησης και κοινοβουλίου με μια σταθερή ε, εύρωστη κυβέρνηση που να μπορεί να προβεί σε λήψη μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, για τη συζήτηση στο G20, στο Brisbane. Ο φορός ο Πρόεδρος Πούτιν έλαβε σαφέστατα μηνύματα από όλους τους ηγέτες που παρίσταντο εσείς πώς ε, εκτιμάτε ότι θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ρωσία και σε αυτό το πλαίσιο πώς ε, θεωρείτε ότι θα κινηθεί ε, η πορεία των πρωτοκόλων και του Μίνσκ Όπως αναφέρατε και εσείς υπάρχουν κάποια ζητήματα με την υλοποίηση των πρωτοκόλων το τελευταίο που αναφέρατε και εσείς ότι σήμερα το πρωί με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυρία Μογγερίνη ε, υπεγράψατε τη συμφωνία ε, για την ε, αποστολή για την μεταρρύθμιση του τομέα πολιτικής προστασίας. Μερικές λεπτομέρειε ακόμα μπορείτε από πλευρά κυβέρνησή σα και να είστε βέβαιο ότι υπάρχει ευρία στήριξη προ εσά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Κυρία Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Πολύ ωραία τα όσα μας είπατε. Εκτιμώ επίσης ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφει. Πολύ θετικό και αυτό. Θα ήθελα να μας πείτε πώς εσείς χειρίζετε τις πολύ κρίσιμες μεταρρυθμίσεις του συστήματος δικαιοσύνης, ε, ε, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτών. και πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά και την ε, πάλι κατά της διαφθοράς. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμεσμάκερ και από τη δική μου πολιτική ομάδα. Κύριε Κλίμκιν, σας καλωσορίζουμε θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως και η δική μας ομάδα σας δίνει την αμέριστη στήριξή τη, Δύο ερωτήματα. Τις τελευταίες ημέρε και ώρες ακούσαμε πολλές ε, δηλώσει, διαβάσαμε πολλές συνεντεύξει, όπου την ρίχνει το φταίξιμο για την ε, κλιμάκωση της κατάστασης στο Κίεβο ενώ υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την κλιμάκωση από ρωσικής πλευράς ε, και πολύ φοβούμαστε ότι θα υπάρχει και ένας φόβος μάλλον για την ε, επανάληψη του περιστατικού της ε, Κρυμαίας. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει πραγματική κατάπαυση του πυρός χωρίς να υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση. Και δεύτερον, ο Πούτιν επίσης άλλη συνέντευξη ανέφερε, υπήρξε μια επένοιξη ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια λύση για την για την κρίση. Εσείς αναφερθήκατε στον όρο «αποκέντρωση». Ο την μιλά για αποκέντρωση και περιφερειοποίηση ως συνώνυμο ε, αυτής της αποκέντρωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, πολλά ομοσπονδιακά κράτη και η Γερμανία αλλά και το δικό μου κράτος, ε, το Βέλγιο, είναι ομοσπονδιακό κράτος. Εσείς πώς ερμηνεύετε ακριβώς αυτή την έννοια της αποκέντρωσης στη χώρα σας, decentralization υπάρχουν, θεωρείται, διαφορές ε, μεταξύ αποκέντρωσης και περιφερειοποίησης ή άλλων όρων. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Ο κύριος ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Εκτιμώ ιδιαίτερως ε, το ανοιχτό σας πνεύμα και την ε, πολύ αυτή λεπτομερή εισήγηση που κάνατε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Το ερώτημά μου αφορά κυρίως ε, ε, την πρόσφατη αύξηση των ε, παραβιάσεων ανθρωπιστικών δικαιωμάτων στις κατεχόμενες περιοχές από τη ρωσική πλευρά της Ουκρανίας, όπως η Κρυμαία. Κύριε Υπουργέ, σε πολλές περιπτώσεις ακούσαμε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις εκφοβισμού και παρενόχλησης των πολιτών της Κρυμαίας που δείχνουν το θάρρος να αντισταθούν στις ρωσικές ενέργειες στην Κρυμαία. Και ως πολίτες της Ουκρανίας προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους βάσει του Ουκρανικού Συντάγματος. Τέτοια περιστατικά ε, ήταν ιδιαίτερα, ε, τέτοιες ενέργειες ε, παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα εναντίον των ταρτάρων, ταρτάρων. Το 2015 είχε προσταθεί ως ε, προθεσμία ε, για να επανεγραφούν τα ουκρανικά ε, μέσα μαζικής ενημέρωσης της Κρυμαίας ως ρωσικά. Ποια είναι η δική σας γνώμη για την κατάσταση στην Κρυμαία και τι πρέπει να γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προβάλλουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα και να προστατεύσουμε τους πολίτες να σαβαστούμε τις διεθνείς δεσμεύσεις ε, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι πλευρέ και η ρωσική διοίκηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας ανακοίνωσε ότι με προεδρικό διάταγμα αναστέλει και τερματίζει όλες τις κυβερνητικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες περιοχές της Ουκρανίας. Δραστηριότητες όμως που χαρακτηρίζουν την κυριαρχία ενός κράτους σε μια περιοχή. Η συνέπειε για τον πληθυσμό των περιοχών αυτών που έχει υποφέρει τα πάντα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπω γνωρίζετε, θα είναι άμεσε και τραγικέ. Αυτό το παραδέχεστε και σπέβδεται να εξαγγείλετε ότι οι πόροι που θα εξοικονομηθούν από την κίνηση αυτή θα διατεθούν σαν ανθρωπιστική βοήθεια για την ανθρωπιστική κρίση που η ίδια η κίνησή σα οξύνει. Κύριε Υπουργέ, είναι αυτονόητο ότι η επιβίωση του πληθυσμού των περιοχών αυτών δεν μπορεί να υπάρξει με ανθρωπιστική βοήθεια. Επομένως, ενδέχεται το κενό που αφήνεται να αναπληρωθεί από τις όποιες αρχές των περιοχών αυτών, οι οποίες θα επιχειρήσουν να βρουν διεθνή πολιτικά και οικονομικά στηρίγματα. Αυτό αποτελεί μια de facto αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης, παράγοντας μάλιστα που προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ένταση από αυτή που διατείνεστε ότι προσπαθείτε να αποφύγετε με τη διατήρηση της εκεχηρίας. Πείτε μου σας παρακαλώ, σε αυτή την εξέλιξη ποια θα είναι η αντίδραση της Ουκρανικής κυβέρνησης και δεύτερον θα συνεχίσετε να αναγνωρίζετε την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Σας ευχαριστώ. One minute. Σε ένα λεπτό, μάλλον τώρα κλείνω κατάλληλο ομιλητών και να μιλάει ο καθένας για ένα λεπτό, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε. Μετά τον πρώτο γύρο συζητήσεων κυρία Χάμ, η πρώτη ερώτηση συνδέεται, αλλά πάει και λίγο παραπέρα από αυτό που ακούστηκαν, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και εκτός των ε, πόλεων που βρίσκονται στο Ντόνιετς και στο Λούγκανσκ, τι μπορεί να κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η παροχή ανθρωπιστικής βιοήθειας σε εκείνους τους ανθρώπους που ε, ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Ντόν και που φοβούνται πώς ε, θα μπορέσουν να επιβιώσουν τον ε, χειμώνα. Για την αποστολή του ΟΑΣΕ ε, φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στην, σε κατάρρευση αυτή η αποστολή. Τι μπορείτε να κάνετε για να σώσουμε αυτό το μηχανισμό που ήταν πολύ σημαντικό; Τι μπορούμε να κάνουμε από τη σκοπιά της δύση για να ε, λειτουργήσει αυτή η αποστολή παρατήρησης. Thank you very much. Mr. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους Ουκρανοί στρατιώτες, παρά τη συμφωνία του Μίνσκ. Ξέρουμε και γιατί είναι μεγάλη συγκέντρωση ε, στρατού από τη ρωσική πλευρά, τάγκ και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού ε, στα σύνορα. Θεωρείτε ότι είναι βιώσιμη η συμφωνία του, του Μίνσκ. Μήπως χρειαζόμαστε κάτι άλλο που να είναι ένα άλλο βήμα, μια άλλη μορφή συμφωνίας που να είναι πιο βιώσιμη. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα ο Τσαριόφ ε, ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά είναι μια κοινή ε, πάλι Ρωσία και Ουκρανίας για να διαμορφωθεί ένα ενιαίο κράτος. Νομίζετε ότι η δυτική εκτίμηση είναι ρεαλιστική? και η ανταπόκριση επαρκής. Αναφέρεται ότι ε, η άρση της, ε, των θεωρήσεων είναι κρίσιμο ζήτημα. Αλλά εάν υπάρξει επίθεση, για... Τι, ποια θα είναι η δική σας ε, απάντηση και ανταπόκριση. Ε, σύντομα το ενδιαφέρον θα στραφεί προς την συμφωνία με το Ιράν. Υπάρχει κίνδυνος η Ρωσία να εκμεταλλευτεί αυτήν ακριβώς τη μεταστροφή του ενδιαφέροντος προς το Ιράν και έτσι ε, εκείνη τη στιγμή να επιτεθεί. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε Κύριο Ζάνι. Όπως ανέφερε ο κύριο Πλάκοβιτ προηγουμένως, υπάρχει σε μια ομάδα διεθνών παρατηρητών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκλογών και εγώ συμμετείχα σε αυτήν την αντιπροσωπεία και μπορώ ειλικρινά να σα πω ότι μάθαμε πολλά. Υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα τα οποία μένουν ανοιχτά κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον και είναι και ένα ερώτημα προς τον ε, Υπουργό. Τι είδου βοήθεια ή συνδρομή χρειάζεστε για να ε, καλυφθούν οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά τη θέρμανση στην Ουκρανία. Και δεύτερον, τι μπορείτε να μας πείτε για, την, για τις έρευνες ό,τι αφορούν ε, το ε, αεροπορικό δυστύχημα με τις ε, αερογραμμές της Malaysian. Γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ο κύριος Βαν και εγώ θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα για τις Malaysian Airlines και τι έχει συμβεί, αν έχετε περαιτέρω πληροφορίες και βέβαια το κύριο ζήτημα είναι η ε, ενεργειακή συμφωνία που έγινε μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θα σταθεί. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει ε, συμφωνία ειρήνης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα ακόμα για την ενεργειακή συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εδώ συζητήσαμε πολύ για τη χώρα σας και θεωρώ πραγματικά τη ε, μεταφορά εξουσίας ε, μετά από τις εκλογές ε, για αυτό τον αδικαιολόγητο πόλεμο. Αυτές οι συζητήσεις, αυτό το οποίο εξετάσαμε είναι ο ρόλος της Ρωσίας. Για το πρόβλημα δεν είναι η Ουκρανία. Θα είμαι ειλικρινής. Θα σας πω μερικά πράγματα εγώ που δεν θα ακούσετε από άλλους που σας κολακεύουν στις ε, Βρυξέλλες και στη Ουάσιγκτον λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για να βελτιωθεί η οικονομία σας ή η κατάσταση στην Ουκρανία. Δυστυχώς είναι ενδιαφέρουσα η Ουκρανία γιατί είναι ένα εργαλείο, ένα αντικείμενο χειραγωγήσιμο μέσα στο νέο ψυχρό πόλεμο που θέλουν πολύ να ε, προχωρήσει. Είναι, αν θέλετε, ένα ε, στη σκακέρα παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο η Ουκρανία. Ελπίζω ότι δεν θα είναι εργαλείο η κυβέρνησή σας και θα καταβάλει προσπάθειες να βρει λύση για όλους τους Ουκρανούς. Μια ομοσπονδιακή λύση που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ότι εδώ μεταξύ μας υπάρχουν ναι, πολλοί φίλοι της Ουκρανίας. Δύο ερωτήματα. Την περασμένη εβδομάδα διάβασα ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός ε, στο Εθνικό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η Γαλλία είναι κυρίαρχο κράτος που κάνει και αντίστοιχες, ε, παίρνει αποφάσεις. Θα συνεχίσει, θα προχωρήσει στην ε, παροχή των Μιστράλ παρά το πολιτικό κλίμα. Τι έχετε εσείς να απαντήσετε στον Γάλλο ε, Πρωθυπουργό. Και κάτι άλλο. Πολλέ πολιτικέ προσωπικότητε στην Ουκρανία θα προτιμούσαν να γίνουν ειρηνευτικέ ε, συζητήσει στο πλαίσιο τη ε, Γενέβη ε, και με παρουσία των ΗΠΑ, όχι με την σύνθεση του Μίνσκ. Και ένα συνάδελφο προηγουμένω ανέφερε. Θεωρείτε ότι η κατάψευση του πυρό, αυτή η ανακοχή είναι επιχειρησιακή ή τέλο πάντων λειτουργεί. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Παρατηρώντας την κατάσταση στην Ουκρανία, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση για μένα. Είναι ανησυχητική επειδή έγιναν εκλογές όπου δεν επρόκειτο μόνο για την εξουσία, αλλά σε διοικητικό επίπεδο, όπως μπορεί να γίνει σε μια χώρα, σε ομαλές καταστάσεις. Στην Ουκρανία όμως κάνουμε λόγο για κάποιες εκλογές σε μια χώρα σε κατάσταση πολέμου. Και σε αυτή τη χώρα σε κατάσταση πολέμου το μισό, το ίμιση του πληθυσμού έμεινε στα σπίτια του και δεν ψήφισε. Και όταν γίνεται λόγος για 80% λέει των Ουκρανών που υπερψήφισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 52% ήταν όσοι συμμετείχαν και στην Ανατολική Ουκρανία μόνο 41% συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κυβέρνησης ιδιαίτερα ευάλωτης, διότι το έθνος δεν ανταποκρίθηκε σε μια στιγμή ιδιαίτερης έντασης ε, που επρόκειτο για την ίδια την επιβίωση της χώρας. Πώς θεωρείτε εσείς ε, ότι με τόσο το χαρακτήρα η κυβέρνηση της Ουκρανίας με τέτοια αποχή των ψηφοφόρων μπορεί να αναλάβει στεναρή δράση υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ της ίδιας της χώρας. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Είναι εξαιρετικά σημαντική παρουσία σας εδώ σήμερα και να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με την Ουκρανία. Θέλουμε να έχουμε ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν, εκτιμούμε όλες ε, τις ε, σχέσεις που έχουμε και μεταξύ πρεσβειών. Εγώ ε, ήμουν παρατηρητής ε, και παρακολούθησα μάλλον τις εκλογές στην Ουκρανία και στην Οδυσσό. Εσείς τονίζετε πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η στήριξη. Πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχουν, ε, να λάβουν χώρα αυτές οι σχέσεις. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο σύνδεσης με τις Βρυξέλλες ή ένας υπεύθυνο εκπρόσωπος. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης που προέκυψε μετά από αυτές τις εκλογές και αναφέρατε αρχικά την καταπολέμηση της διαφοράς. Τι έχετε να πείτε για τις πληροφορίες που λένε ότι υπήρξε χρηματοδότηση από το Παλαμένσκι για την ε, πολιτική εκστρατεία ε, του Γιατσενιούκ the Ευχαριστώ πολύ για τις πολλές και πολύ καλές ερωτήσεις. Νομίζω ότι θα χρειαστώ κάποιες ώρες για να τις απαντήσω όλες λεπτομερώς. Αλλά ας ξεκινήσω με τις πιο σημαντικές ερωτήσεις. προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις μαζί, αλλά χωρίς να χάσουμε καθόλου από την ουσία. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, για, για το σχηματισμό της ε, κυβέρνησης ε, σχηματισμού και αν ε, θα συμμετάσχουν όλα τα μεγάλα κόμματα και τα πέντε φιλοευρωπαϊκά κόμματα συμμετέχουν στην διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης και έχουν τονίσει την δέσμευσή τους. Συμμετέχουν όλα αυτά τα κόμματα, τα φιλοευρωπαϊκά, ε, στην σύνταξη της ε, συμφωνίας. Ε, τώρα, αν θα συμμετάσχουν στην κυβέρνηση ή απλά θα στηρίζουν την κυβέρνηση, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή αλλά το σχέδιο συμφωνίας ε, κυβέρνησης ε, συνασπισμού ε, υποστηρίζεται και από τα πέντε φύρο-ευρωπαϊκά κόμματα. Όσον αφορά την κατάσταση στο Brisbane, πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ποιο, πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι το, το, το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από τις ρωσικές ενέργειες. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την γεωπολιτική αντίληψη του τι συμβαίνει. Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό. Και σκοπός είναι με κάποιον τρόπο η Ρωσία να ελέγχει την Ουκρανία, να μην ε, προχωρήσει στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η Ουκρανία και φυσικά υπάρχουν και διάφορες, ε, κάποιοι διάφοροι συναισθηματισμοί και διάφορες μεταφυσικές προσεγγίσεις, παράλογες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε τον Τόνιας και τον Λούγκανς είναι πρώτα απ' όλα να αναλάβουμε ξεκάθαρες δράσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί ήδη στο Μίνσκ όσον αφορά την ε, διαχωριστική γραμμή, την απόσυρση των στρατευμάτων και την, ε, να καταβληθούν προσπάθειες αρχικά να περιοριστούν και στη συνέχεια να ε, εξαλειφθούν οι περιπτώσεις παραβίασης της κατάπαυσης ε, πυρός. Αν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να μιλούμε για οποιαδήποτε συνεννόηση, για οποιαδήποτε συμφωνία. Και ενέργειες όπως αυτές οι ψευδοεκλογές που έγιναν στις 2 Νοεμβρίου δεν ε, βοηθούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν το σωστό μείγμα. Αλλά και πάλι δεν περιμένω θετικές εξελίξεις. Περιμένω ότι θα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία περαιτέρω αποκλιμάκωσης και γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προσδοκίες μας από την αποστολή της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, αναμόρφωση του συστήματος πολιτικής προστασίας μας. Πρώτα απ' όλα, στη βάση των όσων έχουν ήδη επιτευχθεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα ε, στα νέα κράτη-μέλη, όσον αφορά την επεξεργασία μιας αντίληψης για την αναμόρφωση των αστυνομικών δυνάμεων του συστήματος δικαιοσύνης των βασικών ε, τομέων του, τομέ, του συστήματος πολιτικής προστασίας την επεξεργασία των νομοθετικών πράξεων που χρειάζονται, που απαιτούνται σε αυτούς τους τομείς και στη συνέχεια στην υλοποίηση και την ε, εξέταση των ε, πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Οπότε όλα αυτά συνδέονται με την αναμόρφωση του συστήματος πολιτικής προστασίας και νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον αυτή είναι ε, η μόνη ε, λογική προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσει η αποστολή. Όσον αφορά την, ε, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος έχουμε ένα πακέτο νομοθεσίας κατά της διαφθοράς που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και θα αρχίσει η εφαρμογή αυτού του πακέτου στις αρχές της Άνοιξης γιατί θα πρέπει να προετοιμαστούμε και θεσμικά για την επιβολή, για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Στη βάση ενός προτύπου που εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται φυσιολογικό θα χρειαστεί να δημιουργηθούν ειδικέ μονάδες σε όλη τη χώρα και ειδικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, αλλά για μένα η βασική μεταρρύθμιση, η πραγματική μεταρρύθμιση δεν θα προέλθει από την νομοθεσία, αλλά από το να δημιουργηθεί η αίσθηση στους Ουκρανούς ότι η, η νοοτροπία των δωροδοκιών εξαφανίζεται βαθμιαία για, το, για τη μεταρρύθμιση στο δικαστικό σύστημα. Ε, αποτελούν ε, μάλλον το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ε, μελλοντική συμφωνίας για, την, το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Έχουν ήδη συμφωνηθεί κατευθύνσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από τη δική μας πλευρά στη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο βασικός άξονας των μεταρρυθμίσεων είναι η αναμόρφωση του συστήματος δικαστηρίων στην Ουκρανία διότι εκεί εντοπιζόταν η πηγή ε, πολλών προβλημάτων και για την κοινωνία και για το επιχειρηματικό κλίμα. Ποιος, τώρα, ποιος, ποιος ε, παραβίασε την, ανα, την κατάπαυση πυρός. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το, που το απευθύνουμε και εμείς 20-30 φορές, το, το, δεχόμαστε και εμείς 20-30 φορές τη μέρα. Και τώρα που υπάρχει η αποστολή του ΟΑΕΣΕ, έχουμε περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες περιοχές που προσπαθούν να παρακολουθούν και να ε, ε, επαληθεύουν την ε, κατάσταση επιτόπου. Υπάρχουν μη επανδρομένα αεροσκάφη του ΟΑΕΣΕ. Δυστυχώς κάποια από αυτά καταστράφηκαν από εξοπλισμό παρεμβολών της Ρωσίας καλέσαμε ε, την αποστολή του ΟΑΕΣΕ να παράσχει ασφάλεια και προστασία για τους παρατηρητές μέσω οχημάτων τεθωρακισμένων και για μένα ε, ε, η αποστολή 500 ατόμων στο άμεσο μέλλον θα είναι ο μόνος τρόπος για να επιβάλλουμε την κατάφαση πυρός και να ελέγξουμε την κατάσταση στα ουγρανικά σύνορα. Για την αποκέντρωση και την περιφερειοποίηση, ε, η απάντηση είναι σαφής. Δεν μιλούμε εδώ για χρήση κάποιας ορολογίας, μιλάμε για την ουσία. Φυσικά η Ουκρανία είναι μια χώρα όπου μιλούνται διάφορες διάλεκτοι, όπου υπάρχουν, υπάρχουν διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες, αλλά στο πλαίσιο των ε, πρόσφατων ιστορικών εξελίξεων η ε, Ουκρανία... Ε, στην Ουκρανία ενισχύθηκε το, το αίσθημα της ενότητας και η αποκέντρηση αυτή δεν έχει σκοπό να διασφαλίσει μόνο την ποικιλομορφία αλλά να ε, εξασφαλιστεί η, η οικονομική πολιτική και η πολιτική για την αστρατιωτική ε, ασφάλεια ώστε να παραμείνουμε στο δρόμο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των μεταρρυθμίσεων και της επιβολής του κράτους δικαίου. Οπότε δεν θα δεχθούμε αυτή την ομοσπονδιοποίηση γιατί θέλουν, στόχος είναι να μας κάνουν να αποκλίνουμε από την ευρωπαϊκή πορεία. Άρα δεν μιλούμε για απλή ε, χρήση ορολογίας αλλά μιλούμε για την ε, παροχή ε, περισσότερων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες με την έννοια του να δοθούν περισσότερες ε, ευκαιρίες στις περιφέρειες για να αναλάβουν περισσότερες ε, πρωτοβουλίες. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κρυμαία. Προσπαθώ να θέτω αυτό το ζήτημα σχεδόν κάθε μέρα, διότι η κατάσταση είναι αποκρουστική. Κάθε εβδομάδα ακούμε ε, απίστευτα νέα από την Κρυμαία για την εξαφάνιση ανθρώπων, ιδιαίτερα Τατάρων, της Κρυμαίας και κάποιες μέρες αργότερα κάθε φορά ε, ανεβρίσκονται τα πτώματα των ανθρώπων αυτό. Οι, άνθρωποι ζουν ε, υπό καθεστώς συνεχούς τρομοκρατίας πίεσης και χωρίς να είναι σε θέση να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα. Και για μένα ένα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά θέματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Συμβούλιο της Ευρώπης και για τον ΟΑΣΕ η αποτελεσματική παρακολούθηση της ε, κατάστασης επιτόμου. Και το δικό μου μήνυμα είναι το εξής. Η κατάσταση στην Κρυμαία έχει αλλάξει από έναν φίλο μου που εξακολουθεί να ζει στην Κρυμαία γιατί έχει πολύ μεγάλους σε ηλικία γονείς και δεν μπορεί να τους εγκαταλείψει, μου έστειλε ε, μια φωτογραφία ε, που απεικονίζει ένα σύνθημα στη, Σεβαστού, στη Συμφερούπολη. άνοιξη της Κρυμαίας. Τι θα γίνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Οι άνθρωποι είναι απογοητευμένοι διότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν λάβει πάρα πολύ ψηλούς μισθούς από τους ε, Ρώσους αλλά άλλοι όπως οι Τατάροι της Κρυμαίας ε, έχουν αφηθεί στην τύχη τους. Ο τουρισμός ε, στην Κρυμαία έχει καταρρεύσει. Μια περιοχή όπου το, τα δύο τρίτα των ανθρώπων εξαρτώνταν από τον τουρισμό. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας, αλλά θα πρέπει ε, επίσης να αποστείλουμε και ένα σαφές μήνυμα για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για να προστατευτούν οι Τατάροι της Κρυμαίας Και πρότασή μου είναι να ε, προσκαλέσετε εδώ σε συνεδρίαση της ΑΦΕΤ τους ηγέτες των Τατάρων για να ε, έχετε και μια άμεση επικοινωνία μαζί τους με τον κύριο Τζέμιλοφ ή με τον κύριο Τζουμπάεφ που υπέφεραν και στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης και τώρα ξανά υποφέρουν λόγω της ρωσικής κατοχής. Για την ανθρωπιστική βοήθεια έγινε μια παρακήρυξη κρίσιμη σημασία γιατί τους τελευταίους μήνες προσπαθούμε να οργανώσουμε τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Ντόνιασκ και το Λούγκανσκ να συγκεντρώσουμε αυτοκινητοπομπές να αποστείλουμε εκεί, να εξασφαλίσουμε τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε μόνο ρωσικές αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν κάτι, δεν ξέρουμε τι όμως. Πριν από μια εβδομάδα έγινε μια ακόμη προσπάθεια για αποστολή, για παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες του Ντόγιανσκ που απέτυχε όμως λόγω της παρουσίας των στρατοτών διότι οι τρομοκράτες υπό τον έλεγχο των Ρώσων απλώς και μόνο δεν μας επιτρέπουν να παραδώσουμε ή εσδήποτε μορφής ανθρωπιστική βοήθεια φοβόμενοι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την οτροπία, τη στάση, την ε, στις θέσεις των πολιτών εναντί και άρα την επιλογή του ποιο θα πρέπει να διαχειρίζεται αυτέ τι περιοχέ. Όμω εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και έξω από τα κατεχόμενα από του τρομοκράτε εδάφη. Υπ' αυτή τη ενία οι διμερεί επαφές και η διεθνής υποστήριξη θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο πολύ αποτελεσματικό με τους παρατηρητές που έχουν πάει και από τη ρωσική ε, πλευρά σε δύο, σε δύο σημεία ελέγχου όπου εκεί πρέπει να πω ότι δεν ήταν αποτελεσματική για το λόγο ότι δεν επιτρέπουν απλά και μόνο οι Ρώσοι δεν έχουν διάθεση να επιτρέψουν στους διεθνείς παρατηρητές τον, ε, την παρακολούθηση του ελέγχου των συνόρων. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί οι παρατηρητές, παρακολουθούν τα πράγματα σε αυτά τα δύο σημεία ελέγχου, αλλά έστω και έτσι μπόρεσαν να διαπιστώσουν πολλά πράγματα. Επί παραδείγματι κάποιους που κουβαλούσαν πολύ εξοπλισμό και πυρομαχικά και περνούσαν τα σύνορα, αλλά και περνούσαν και από άλλα σημεία ε, ή από άλλες διαδρομές μεταφέροντας και με φορτικά ακόμη εξοπλισμό. Όλα αυτά βρίσκονται τώρα στον ιστότοπο της αποστολής των παρατηρητών. Μπορούν να αντέξουν ακόμη συμφωνίες του Μίνσκ. Ναι, βεβαίως, εμείς είμαστε ως κράτος απολύτως και απαρέγκλητα προσκολλημένη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ε, παρά μόνο εάν θέλει κανείς βέβαια να ε, οδηγήσει σε κλιμάκωση και ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση την κατάσταση. Μπορούμε για ώρες να κάνουμε υποθέσεις για το ποια θα μπορούσε να είναι μια καταλληλότερη αντίδραση ή κατάλληλη αντίδραση και αν είναι ρεαλιστική η αντίληψη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και να πούμε ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη γραμμή τη, όχι μόνο βέβαια για τι κυρώσει, γιατί οι κυρώσει είναι ένα μέρο και μια όψη μόνο του νομίσματο, σημαντική μένα, αλλά μόνο μία. Πρέπει να καθίσετε όμω απόλυτο σαφέ σε κάθε μορφή επαφή, επικοινωνία, διμερού σχέσεω, ότι η σταθεροποίηση είναι προϋπόθεση για περαιτέρω σχέσεις. Δεν είναι σαφές ακόμη το πώς μπορεί να παγώσει η κατάσταση του Λουγκανσκ και του Ντόνιεσκ και να παραμείνει ως παγωμένη σύγκρουση αντίστοιχη με τις Απχαζίας και τις Πιδοσυνθερίας. Ε, για δε το αεροσκάφος και την κατάρριψή του των μαλαισιανών αερογραμμών ήταν σαφές νομίζω αυτήν την εβδομάδα με την παρουσίαση και την παρουσία εκπροσώπου του εισαγγελέα των κάτω χωρών. Κάναμε πολλές διαβουλεύσεις και προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε κομμάτια, συντρίμια του αεροπλάνου που θα προσφέρουμε στις αρχές των κατοχωρών, τις αγγελικές αρχές. Αυτό είναι βέβαια πολύ δύσκολο γιατί οι τρομοκράτες έχουν κάνει τεράστια ζημιά ήδη. Αλλά πιστεύω και ήταν και η πρωτοβουλία δική μου ότι οφείλουμε να δώσουμε την πρωτοκαθεδρία στους Ολλανδούς φίλους ε, για την έρευνα αυτή είναι σωστό και πολιτικά όσο και δεοντολογικά. Ήταν η σωστή λύση και απόφαση αυτή και πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει εν τέλει σε μια πραγματική διαφανή και αμερόληπτη έκθεση του τι συνέβη, όχι μόνο την ε, ημέρα εκείνη και με την τραγωδία αυτή, αλλά και σε σχέση με τις πηγές της τραγωδίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας βοηθήσει έτσι και να προς, προσαγάγουμε τους υπετίους ενώπιον της δικαιοσύνη και όχι απλώς να αναζητούμε ποιες ήταν οι πραγματικές αιτίε. Το θέμα των ελλείψεων σε θέματα θέρμανσης και παροχή φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει τίποτε. Το απόκριφο ή το απόρριτο σε σχέση με τη συμφωνία για το φυσικό αέριο είναι απόλυτα διαφανή στη διαδικασία. Είναι σημαντικό να επιτύχουμε με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είμαστε σε θέση να αγοράζουμε σχετικά μικρή ποσότητα φυσικού αερίου με τιμή που έχει οριστεί μέσα από τη σύμβαση με προκαταβολή μόνο του τιμήματος. Εάν χρειαζόμαστε δηλαδή ένα δισεκατομμύριο κυβικών μέτρων, μπορούμε να προεξοφλήσουμε ένα δισεκατομμύριο και να πάρουμε ένα δισεκατομμύριο. Εάν χρειαστούμε δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα πληρώσουμε δύο δισεκατομμύρια προκαταβολικά και θα λάβουμε δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αλλά μην ε, παρερμηνεύεται αυτή η συμφωνία. Πρόκειται για την παλιά σύμβαση που πάει μέχρι τα τέλη του Μαρτίου, όχι για τη νέα, για την οποία αναζητούμε πιο σαφεί εικόνε για το πώ μπορούμε να χειριστούμε τα θέματα του φυσικού αερίου. Έχουμε τη διατησία της Στοκχόλμης για το σοβαρό αυτό πρόβλημα και αναμένουμε μια δίκαιη και μερόληπτη απόφαση από τη διατησία αυτή, τη διεθνή διατησία της Στοκχόλμης, βάσει της οποίας θα μπορέσουμε να συνάψουμε μια νέα σύμβαση με πραγματικές δίκαιες τιμές, με βάση τα όσα ορίζει η αγορά, για να, ε, για ε, εφοδιαστούμε σε φυσικό αέριο και στο μέλλον. Κάτι το σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για εμάς, γιατί αφορά την κοινή μας ασφάλεια. Γιατί τα Μιστράλ είναι σαφές, και το είπα και από την αρχή, ότι η παράδοση των Μιστράλ είναι εναντίον κάθε πολιτικής λογικής, εναντίον του κώδικα ε, δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν πραγματοποιηθεί δεν θα πρέπει να υπονομεύει την ασφάλεια, αλλά να οδηγεί στην ενίσχυση της ασφάλειας για τέτοια επιλογή για το μέλλον. Άρα, οι Γάλλοι εταίροι και φίλοι θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα λύση, στοχευμένη για τα Μιστράλ, αλλά πάντως δεν πρέπει να τα παραδώσουν. Διότι εν τέλει μια τέτοια κίνηση υπονομεύει όχι μόνο τη δική μας ασφάλεια, αλλά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι και το μήνυμά μου. Για το φόρματ της Γενέβης, εγώ το υποστηρίζω σαν συσχετισμό και συνομιλίες. Προσπαθώ να προωθήσω μια δεύτερη τέτοια συνάντηση Θέλω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Θέλω να είναι και οι Ηνωμένε Πολιτείε γύρω από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και άρα για μένα αυτή θα είναι και η λύση. Οι Ρώσοι διστάζουν να τη δεχθούν. Αλλά εγώ θα εργαστώ καταπώνητα προς τη λύση αυτή. Η ιδέα ότι μόνο 50% προσήλθαν στην, στην ε, κάλπη, 52% των Ουκρανών ψήφισαν στις εκλογές αυτές. Το αποτέλεσμα όμως είναι σαφές. Μπορεί να σας φαίνεται παράδοξο, αλλά με όλα τα, όλες τις δημοσκοπήσεις που έγιναν, οι Ουκρανοί δήλωσαν ότι είναι σίγουροι για την φιλοευρωπαϊκή επιλογή και στροφή και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ήταν τόσο δε σίγουροι που τελικά δεν πήγαν να ψηφίσουν, ε. έμειναν στα σπίτια τους. Αν διαβάσετε όμως τα αποτελέσματα των εκλογών, όχι μόνο για το Κίεβο ή την Νότια Ουκρανία, και ούτε μόνο στην Ανατολική Ουκρανία. Παντού, παντού είναι πολύ σαφές το αποτέλεσμα και ξεκάθαρη πλειοψηφία υπέρ των κομμάτων που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη περιοχή της Ουκρανίας όπου ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης να κέρδισε στην περίπτωση αυτής της εκλογής. Εγώ προσωπικώς θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συμμετοχή του εκλογικού σώματος στις ε, εκλογές, αλλά νομίζω ότι φτάνουμε πια στα επίπεδα τα ευρωπαϊκά. Ε, και για τις ευρωεκλογές είναι κάτω από το 50% η συμμετοχή. Και για τους Ουκρανούς βέβαια το 52% είναι μεγάλη πρόκληση, γιατί θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά στην πολιτική, στο πολιτικό γίγνεσθε και την αντιπαράθεση στην πολιτική τους πολίτες πώς μπορεί να υπάρχει επαφή με τις ευρωπαϊκές ε, αρχές. Θα υπάρχει ένα σύστημα συντονισμού για την παρακολούθηση και το συντονισμό όλης της ευρωπαϊκής πορείας. Διαφορετικές ιδέες εκφράζονται, όμως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ειδικό γραφείο, γραφείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με πολλούς αρμοδίους που έχουν αναλάβει τον, ε, την κατάρτιση της συμφωνίας και την αναζήτηση στους διάφορους τομείς όπου υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη και τις επαφές αντίστοιχα με, τα ευρωπαϊκά όργανα. Και γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι έχουμε καταστήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δεν την έχουμε υπαγάγει στο, εξωτερικό, στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά σε ε, θέματα εσωτερικά, γιατί θεωρούμε ότι είναι εσωτερικό ζήτημα αυτό το της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας. Για, τα, για τις δαπάνες της προκλογικής εκστρατείας και τους υπενιγμούς ότι μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιους ε, ε, μεγάλο επιχειρηματίες ή ολιγάρχες όπως τους λέμε. Κοιτάξτε, έχει αναλάβει τέτοιου είδους διερεύνηση και μέρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, παρά όμως την διεξοδική έρευνα από δημοσιογράφους δεν έχει προκύψει τίποτα το συγκεκριμένο. Άλλωστε ολόκληρη εκστρατεία έγινε μέσω της τηλεοπτικής οθόνης. Πολύ, λίγο, πολύ λίγες εκδηλώσεις έγιναν έξω από, την, από τον τηλεοπτικό φακό. Άρα όλα έγιναν κατά τρόπο δημοκρατικό και με λιγότερα έξοδα από ό,τι πρέπει. Όλα αυτά νομίζω ότι έχουν και το συμβολισμό τους. Για να κλείνω λοιπόν και ελπίζοντας να έθιξα όλες σας τις, ε, όλους τους προβληματισμούς προσπαθώ να μην ε, συνοψίσω υπερβολικά τα ερωτήματα, τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου μπορώ να σας μιλήσω σήμερα, για την υποστήριξη σας ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε την έκφραση της ευγνωμοσύνης της περιόδου. περιόδους, τη χρειαζόμαστε και ε, οι Ουκρανοί και πάνω απ' όλα για τα θέματα αυτά που έχουν τόσο μεγάλη σημασία για τους Ουκρανούς, την ευρωπαϊκή δηλαδή θεώρηση, την τομεακή ολοκλήρωση, την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης, και όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σε ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας εκθέσατε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και τύχη για τη χώρα σας να είσαστε βέβαιοι ότι δεν θα παρατηρούμε και παρακολουθούμε μόνο, αλλά και τη δημοκρατικά εκλεγήσα κυβέρνηση της Ουκρανίας θα την υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστούμε που προσήλθατε. Συνάδελφοι, το σημείο για τον Καναδά μπορούμε να το επισπεύσουμε, αν συμφωνείτε διότι θα ήθελα να συνοδέψω τον κύριο Υπουργό για μια συνέντευξη τύπου και θα ήθελα σε σχέση με την Γεωργία να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Καναδάς πρώτα. Ο εισηγητής θα λάβει τον λόγο. Charles Τένοκ. έχετε τον λόγο κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Μέσμακα θα το αναλάβει, θα είναι προεδρεύον παρακαλώ.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 Okay, dear colleagues. Εντάξει, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακαλώ τώρα με τις εργασίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων εκείνοι που αποχωρούν. Έχουμε τώρα σε σχέση με το θέμα της ε, ε, συνέντευξης του κυρίου Κλίμκιν ήσυχα να αποχωρήσετε. Περνάμε στο 6 της ημερήσιας διάταξης ε, συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά μεταφορά των ε, στοιχείων δεδομένων ταξιδιωτών εναέριων ε, εταιριών ε. και θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν εσείς κύριε Ντεμέσμακα να λάβετε τον λόγο. Παρακαλώ. Πρέπει να ζητήσω, τον, να ζητήσω συγγνώμη για τον κύριο Τάνοκ που λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να παραστεί. Θα παρουσιάσω εγώ τη γνωμοδότησή του. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή υπενθυμίζεται συχνά η απειλή της παγκόσμιας τρομοκρατίας και σε σχέση με την Ευρώπη και την παγκόσμια κλίμακα αυτού του φαινομένου, το οίκης είναι η τελευταία έκφραση αυτού του φαινομένου. Μην ξεχνάμε ότι 3.000 υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάχονται στη Συρία και το Ιράκ υπό την οίκης καθώς ομιλούμε αυτή τη στιγμή. Υπό αυτό το πλαίσιο για την ασφάλεια θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα προτερήματα αυτής της συμφωνίας με τον Καναδά όπως προτείνεται. Φυσικά έχω συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει οξία αντίδραση σε αυτή τη συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο. Όμως θα ήθελα να προσπαθήσω να ζητήσω να είμαστε πιο ρεαλίστες. Η συμφωνία του 2006 συνεχίζει να εφαρμόζεται και να λειτουργεί και η συμφωνία που συζητούμε σήμερα προσφέρει βελτιωμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά για τους ε, υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιορισμένη περίοδο αποθήκευσης αυτών των στοιχείων που είναι ακρογωνιαίοι λύθη αυτής της ε, συμφωνίας καθώς επίσης και σημαντικούς ε, βαθμούς πρόσβασης, πελασιμότητας και διαδικασιών επανόρθωσης. Υπάρχει συζήτηση και πρόταση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να γίνει μια προσφυγή στο 10, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι έτσι όμως θα έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια ολόκληρα και δεν θα διασφαλιζόταν ένα υψηλό επίπεδο προστασία για του Ευρωπαίου πολίτε για τα προσωπικά του δεδομένα. Φυσικά είναι συζήτηση που πρέπει να διεξαχθεί και να επιληθεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά ζητήθηκε να υπάρξει γνωμοδότηση για αυτή τη συμφωνία υπό του όρου τη εξωτερική πολιτική και των θεμάτων ασφαλεία, που είναι δικέ μα αρμοδιότητε και ως προς αυτά διασφαλίζει τη ζωτική συνεργασία αυτή η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και του Καναδά, εταίρου στο ΝΑΤΟ ο Καναδάς και σύμμαχός μας στην μάχη κατά της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Υπενθυμίζοντας όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Τάνοκ συνιστά ως εισηγητής η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεμέσμακερ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποιος άλλος από τους συναδέλφους, θα ήθελα να λάβει τον λόγο. Εσείς ως κοιόδης εισηγητής από το ΕΛΚΑ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λέει ο Κοβάτσεφ, του συναδέφους για το έργο που επετέλεσαν. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ε, εγκλημάτων είναι χρήσιμη αυτή η συμφωνία στην εργαλειοθήκη μας. Η αποτελεσματική ανταλλαγή στοιχείων όπως και των στοιχείων ταξιδιωτών ήταν χρήσιμο στοιχείο ως προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και είναι ένα χρήσιμο μέσο, ένα χρήσιμο εργαλείο για την δίωξη και την ε, ε, επιβολή κυρώσεων. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τους εταίρους μας όπως τον Καναδά θα έπρεπε κανείς να υπογραμμίσει ότι ο, ο ίδιος βαθμός προσοχής πρέπει να δίνεται και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Έχουν το δικαίωμα οι Ευρωπαίοι πολίτες να ζητούν να υπάρξει διασφάλιση αυτών των δεδομένων και δυνατότητα επανόρθωσης. Και η συμφωνία ευθυγραμμίζεται με την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς εγκλήματος ώστε να διασφαλίζεται η διαβίβαση αυτών των στοιχείων. Έχουμε παρόμοιες συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία και με τον Καναδά από το 2006 όπως προανέφερε ο συνάδελφος. Ζήτησε την τροποποίηση αυτής, αυτής της συμφωνίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτών των συμφωνιών Πράγματι συνέβη αυτό με τη ΣΥΠΑ και έχουμε ένα τροποποιημένο κείμενο και τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο και να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Καναδά. Καμιά φορά δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση όσον αφορά την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που προέρχεται από κάποιες πολιτικές ομάδες. Το να πετύχουμε μια συμφωνία έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα. Μια και ταξιδεύουν Ευρωπαίοι πολίτες ε, στη Μέση Ανατολή και υπάρχει και η εμπλοκή ε, Ευρωπαίων πολιτών ε, στην Ίκης. Δεν αναμένουν οι τρομοκράτες τη δική μας αυτή αναθεώρηση. Πρέπει εμείς τώρα άμεσα να δράσουμε χωρίς καμιά καθυστέρηση. Και τέλος να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο χρόνια στη Βουλγαρία υπήρξε μια τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο του Πύργου, του Μπουργκάζ, όπου από την Αυστραλία και τον Καναδά, αρχικά από τον Λίβανο, υπήρξε αυτή η εμπλοκή τρομοκρατών. Χωρίς ε, την συνεργασία των ε, διοκτικών ε, αρχών δεν θα μπορούσαμε να διακριβώσουμε ποιοι ήταν πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Να το ξαναδείτε, να το ξανασκεφτείτε συνάδελφοι και να πούμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ότι πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο έκθεσης για αυτή τη συμφωνία με τον Καναδά ώστε να μπορέσει να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοβατσέφ. Ήταν σαφέστατη έκκληση στην Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Έχετε τώρα εσείς τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζουμε τον περίπλοκο χαρακτήρα αυτού του προβλήματος, λέει ο κύριος Σασίς. Ε, εδώ είναι ε, μια σύγκρουση αξιών όσον αφορά την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και το θέμα της ε, διασφάλισης της ασφάλειας σε παγκόσμια κλίμακα ιδιαίτερα όσον αφορά Ευρωπαίους. Γνωρίζουμε ότι αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και οποιαδήποτε απόφαση είναι μια απόφαση που πάντα έχει περίπλοκο και σύνθετο χαρακτήρα από τη μία πλευρά έχουμε τις θεμελιώδεις αρχές ε, του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, την διασφάλιση της αυτονομίας, την εγγύηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων για τους πολίτες μας, εδώ με την προστασία δεδομένων και από την άλλη πλευρά μια άλλη αξία που είναι η αξία της ασφάλειας που πρέπει και αυτή να διασφαλιστεί. Και θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες ε, με άλλες περιοχές και άλλες χώρες όπως έχουμε ήδη ε, κάνει. Το θέμα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει καθορίσει επακριβώς την ομοθεσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία προσωπικών δεδομένων το τι θα γίνει δηλαδή σε σχέση με κάθε μια από αυτές τις συμφωνίες. Και έχουμε πρόσφατα απόφαση νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 10, αντίθετα δηλαδή προς κάποιες συμφωνίες που είχαν συναυθεί. Ως προς αυτό θεωρούμε ότι είναι πιο λογικό, πιο συνετό αυτή τη στιγμή να αναμείνουμε, να υπάρξει σαφής νομοθεσία που θα εκπονηθεί σε αυτόν τον τομέα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών, πράγμα που φυσικά πρέπει να γίνει με τον πιο ταχύ, τις ταχύτερες διαδικασίες ε, από την άλλη πλευρά πρέπει αυτή η νομοθεσία να εφαρμόζεται σε συμφωνίες με άλλες χώρες και άλλες περιοχές του κόσμου δεν έχουμε κάποια επικριτική τοποθέτηση όσον αφορά τέτοιες συμφωνίες, αλλά έχουμε αυτή την ανησυχία να υπάρξει η διαφύλαξη κάποιων αρχών που θεωρούμε εμείς ότι είναι συντακτικές αρχές και αξίες ε, του δικού μας πολιτισμικού εγχειρήματος και δεν μπορούν να, να αμφισβητηθούν ή να υπονομευθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί διαφορετικά θα δεχόμαστε να ενταχθούν ε, θέματα στην, ε, στην προσπάθειά μας οι μεγαλύτερες απειλές για παράδειγμα που υπονομεύουν ε, το δικό μας πρότυπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σις. Η κυρία Νέιτς τώρα θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ε, παίρνω τη θέση της ε, κυρίας Μαρίτης Χάκε που είναι σκιώδης ε, για αυτή την γνωμοδότηση και δυστυχώς δεν είναι εδώ. Θα εκφέρω λοιπόν τη δική της γνώμη με την οποία δεν συμφωνώ απαραίτητα. Η κυρία Σχάκε έχει υπεβάλει τροπολογία με την οποία ζητά από το Κοινοβούλιο να μην συνενέσει, να μην εγκρίνει αυτόν τον κανονισμό για λόγους ε, που νομίζω έχει εξηγήσει και σε προηγούμενες συζητήσεις για παρόμοιους, ε, παρόμοιες ε, με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. σχετικά με προβληματισμούς ό,τι αφορά την καταλληλότητα της νομικής βάσης, την αναγκαιότητα τέτοιας μαζικής συλλογή δεδομένων, την αναλογικότητα των κανονισμών, το εύρος των σκοπών που μπορεί να επικληθεί κάποιος για τη συλλογή τέτοιων δεδομένων και κατά πόσο επαρκούν οι δυνατότητες δικαστικής εποπτείας γιατί εκείνη θεωρεί ότι σε όλα αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια. Γι' αυτό και συστήνει αρνητική ψήφο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, το 2009 στο 2012 παρακολουθούμε τι έχει συμβεί με ε, την ε, τρομοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι επίγον το ζήτημα και υπάρχει αναγκαιότητα να δράσουμε για να προστατεύσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Η τρομοκρατία αναπτύσσεται και γεωγραφικά και τεχνολογικά. Έχει περισσότερα μέσα δράσης και εμεί δεν γίνεται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ε, ακούω να λένε συνάδελφοι να μιλάνε για προβλήματα νομικά ε, και για αρχές προφύλαξης, απαραίτητο, αλλά αν υπάρξουν σωματικές επιθέσεις τρομοκρατικές, τι θα πούμε στις οικογένειες των θυμάτων. Θα τους πούμε ότι ναι, ξέρετε, καλά τα λέτε, αλλά εμείς ε, έπρεπε να τα συζητήσουμε και να δούμε τα νομικά πριν αποφασίσουμε. μιλάμε για την τρομοκρατία, αλλά και την αύξηση της κινητικότητας και της ευελιξίας των τρομοκρατικών ομάδων. Κινητικότητα, δηλαδή τη δυνατότητά τους να αξιοποιούν όλα τα μειονεκτήματα, τα ευάλωτα σημεία της νομοθεσίας μας ε, και της, ε, της σύναψης σχέσεων, ή μάλλον εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά με τις χώρες με τις οποίες εμείς δεν έχουμε τέτοιες συμφωνίες. Κι όμως εδώ αυτή η πρόταση μας επιτρέπει ακριβώς να ενεργήσουμε και να πούμε ότι θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες χώρες με τις οποίες θα έχουμε τέτοια συμφωνία. Και αφετέρου αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα της ευελιξίας τους, γιατί εφόσον ε, εμείς ενεργούμε μόνο σε κάποιες χώρες, εκείνοι θα έχουν τη δυνατότητα να περνάνε από αλλού. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το ψήφισμα είναι εξαιρετικά ε, ισορροπημένο και υπάρχει πραγματική αναγκαιότητα και εμείς φέρουμε πολύ σημαντική ευθύνη εάν αφήσουμε ανοιχτές διόδους για τους τρομοκράτες. Um, Η ε, κυρία Γκόμες, ως μέλος και της Επιτροπής ε, ΛΥΒΕ και έχοντας γνώση και των συζητήσεων που γίνονται εκεί, παρότι ξέρω ότι στην περίπτωση της συμφωνίας με τον Καναδά έχουν επιληθεί κάποια ζητήματα που είχαμε με τη ΣΥΠΑ, παραμένουν κάποια ζητήματα συνοχής. Και διατύπωση ή διάρθρωσης. Δεν μπορούμε να δώσουμε προηγούμενο όταν ακόμα δεν έχουμε επιλύσει σημαντικά στοιχεία μεταξύ μας. Δεν έχουμε στην Ευρώπη, για παράδειγμα, ε, τέτοιο σύστημα συλλογής δεδομένων ταξιδιωτών του PNR γίνεται χαμός. Η κάθε, κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική συμφωνία με επιμέρους χώρες και τα πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ε, μπερδεμένα. Ε, συγγνώμη, αλλά αυτό το επιχείρημα για την δρομοκρατία δεν νομίζω ότι πείθει και πολύ τους πολίτες μας. Χθε ήμουν στη χώρα μου σε μια συνεδρίαση με πολλούς προσκεκλημένου και τον κύριο Ασάντζ μέσω τηλεδιάσκεψη και μπορώ να σα πω ότι αν δεν τα πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά και έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και αντιμετώπιση, πάντα σεβόμενοι τις αρχές μας, αλλά σε συνδυασμό και με την ανάγκη για ασφάλεια, τότε πραγματικά δεν υπηρετούμε τα συμφέροντα ούτε της Ευρώπης, ούτε των πολιτών μας και της προστασίας τους. Γι' αυτό καλό είναι να ακολουθήσουμε ε, τη γνώμη ε, του κυρίου Ασή και τη κυρία Τεσχάκη. Γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε συνοχή. Συνοχή και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Πρέπει να συνεργαστούμε με του συναδέλφου από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και να γίνει μια πραγματική ανταλλαγή ε, απόψεων και να ακολουθήσουμε στρατηγική προσέγγιση. Να μην έχουμε ένα συνοθήλευμα διαφορετικών γνώμεων. Ah Αν είναι πραγματικά απαραίτητο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, τότε αυτό μπορεί να, γίνει και με μια ε, συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία που εδώ έχει καταρτιστεί δεν εξυπηρετεί την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γι' αυτό τον σκοπό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να καλέσω όλους να ε, εξετάσουν πολύ, με πολύ κριτικό μάτι την προτινόμενη συμφωνία. Πρόεδρος. Για την συμφωνία σύνδεσης με τη Γεωργία. Κύριε Ισηγητά, ε, θα πρότεινα η συζήτηση για το 4 και το 5 να γίνει από κοινού. Έχετε κάποια παρατήρηση? Δεν υπάρχει ούτε από τους συναδέλφους, οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ποιος είναι Ψηφίζουμε για το σχέδιο σύστασης, για, την, ε, για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και ε, ξεκινά. Ε, αν θέλετε τον λόγο. Ε, και είπατε όχι. Κύριε Σιγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ε, δεν κατάλαβα ότι Μα είχατε πει να πάρουμε το λόγο. Συνάδελφοι, αρχικά θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω του ασκιώδει εισηγητέ για την ε, το ομαδικό πνεύμα, το πνεύμα συμβασμού και πριν ψηφίσουμε θα ήθελα να πω τα εξή. Α στηρίξουμε την ευρωπαϊκή επιλογή τη Γεωργία. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία. Die Abstimmung ist πέρας angenommen τώρα. Εγκρίθηκε 46 υπέρ, 2 εναντίον, 3 αποχές. Θερμά συγχαρητήρια. Και συγχαίρουμε και τη Γεωργία εξίσου. Με μια ισχυρή εντολή λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε προς επικύρωση την οποία θα συστήσουμε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και περνάμε στο ψήφισμα. Για το ψήφισμα θέλουν κάποιοι να παρέμβουν. Δεν επιθυμεί να παρέμβει κάποιος. Ψηφίζουμε λοιπόν. 33 υπέρ. 35 διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ. Τροπολογία 35. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 36. Πέρας ψηφοφορίας. 20-31 το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 43 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 42. Πρέπει και αυτή να την ψηφίσουμε. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 42 λοιπόν. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 23-28 το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Περνάμε στην 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 47 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 47. Άρχεται. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. ψηφοφορία ψηφοφορίας τώρα. 26-23 εγκρίθηκε λοιπόν. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 54 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 54, άρχεται η ψηφοφορία. Η 54, έτσι. Πέρας ψηφοφορίας, 31-20, απορρίφθηκε. Η 54 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 υπέρ κατά 56 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 75 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 75 άρχεται πέρας ψηφοφορίας 25-25 η ισοψηφία απορρίφθηκε. Μπορούμε να σταματήσουμε τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πτερίγων του ΕΛΚ. Να πάψουν οι συζητήσεις παρακαλώ. Εβδομήντα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 89 υπέρ Όχι λέει ο πρόεδρος. 87 λοιπόν. 87 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 87. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 35-18. Απορρίφθηκε. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε φυσικά διορθώνει ο πρόεδρος. 35-18 εγκρίθηκε. Αυτή ήταν 87. 88 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι φιλελεύθεροι ήθελαν να παρέμβουν πριν από το συμβιβασμό 4, πριν ψηφίσουμε τη συμβιβαστική 4. Παρακαλώ λοιπόν οι φιλελεύθεροι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μόνο για να υπάρξει μια επανόρθωση, μια μικρή τροποποίηση ως προς το ότι στην παράγραφο στην οποία αναφερόμαστε στη Ρωσία ως the main actor, ο κύριος εμπλεκόμενος, να αλλάξει ως ένα σημαντικός εμπλεκόμενος. Και έχει νόημα αυτό να μην ε, αναγνωρίσουμε τον κύριο, κυριότερο ρόλο με μια τέτοια λειτουργία στρατηγικά αποφασιστικού χαρακτήρα από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να το αλλάξουμε λοιπόν το as the main actor ως ο κύριος εμπλεκόμενος να το αλλάξουμε σε έναν σημαντικό εμπλεκόμενο. Αυτό να γίνει. Έχει νόημα αυτό. Υπάρχει αντίρρηση. Αν όχι γίνεται δεκτή η τροποποίηση. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 4 με αυτή τη διατύπωση. Ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, Συμβιβασμός 4 λέμε, compromise 4. Έγινε μια τροποποίηση προηγούμενα, εντάξει, και την ψηφίζουμε με αυτή την τροποποίηση. Αντί ο κύριος εμπλεκόμενος, ένας σημαντικός εμπλεκόμενος. Ιδιαίτερα το ΕΛΚ θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την πρόταση, έτσι. Ωραία, λοιπόν, ψηφίζουμε και πάλι το συμβιβασμό 4, υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 116 που βρίσκεται εδώ. 116 λοιπόν υπέρ. 116 δεκαέξι, ένα παρακαλώ. 1-1-6 Μετά την 122 τροπολογία, εντάξει, στη σειρά. Το βρήκα, ε, αλλά ήταν δύσκολο με αυτόν τον κατάλογο. Εν πάση περιπτώσει. 116 τροπολογία. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 129. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 130 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε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 Πέρας ψηφοφορίας. 29-23 εγκρίθηκαν λοιπόν. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 η 13 εγκρίθηκε πιο πριν. Μάλιστα. Περνάμε στην 22. 21, 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίθηκε. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ 6, 6 υπέρ λοιπόν. Κατά Θέμα συμμετοχής των μελών. Δηλαδή ποιος θα ψηφίσει για τους χριστιανοδημοκράτες, ένας όλος και όλος, τι γίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε, ψηφίζουμε την εξι άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 23-31. Έγινε σφάλμα τότε λοιπόν. Λοιπόν, για να το δούμε. Ναι, το γνωρίζω αυτό λέει ο Πρόεδρος. Στην παράγραφο 3 έκανα ένα σφάλμα λέει ο Πρόεδρος. Όταν είχαμε τη 43 και απορρίφθηκε, στη συνέχεια η 44 τροπολογία θα έπρεπε να ψηφιστεί. Δεν το έκανα, πήγαμε στη 45. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να επαναλάβουμε, να καλύψουμε αυτή την ανάγκη αυτής της ψηφοφορίας. Ποιοι είναι υπέρ της 44, ο Στρεβίτσιος και τα λοιπά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε η 44. Και το ίδιο λοιπόν σε σχέση με την 45. 45. Όχι, όχι. 45 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ωραία, την 7 την είχαμε, να ψηφίσουμε την 7 λοιπόν, όσοι θέλουν να ψηφίσουν, υπέρ της 7 λοιπόν ή κατά, κατά αποχές εγκρίθηκε η 7. Περνάμε τώρα αμπλόκ στο σύνολό τους στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε όλες συνολικά υπέρ αυτών. Κατά αποχές εγκρίθηκαν λοιπόν. Και περνάμε στη συνέχεια στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ψηφοφορία επί του κειμένου ε, της έκθεσης, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ονομαστική, με ονομαστική κλίση. 49 υπέρ 3 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια θερμά προς τον εισηγητή, κύριο Μαμίκινς. Πέρα συνεδριάσεως.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 Dear colleagues, the break will last another four or five minutes before Mingarelli comes, so you can feel free to have a break. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πέντε λεπτών μέχρι να έρθει ο κύριος Μιγκαρέλη. Bon, chers collègues, je vous prie de recommencer notre Μπορούμε να ξανασυνεχίσουμε με το σημείο 7 στην μέση διάταξη, το σημείο ενημέρωση με τον κύριο Ιγκμαν Τζαρελή από, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, αρμόδιο για θέματα Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Αραβική Χερσονήσου, Ιράν, Ιράκ. Θα μα ενημερώσει για τι πιο πρόσφατε εξελίξει στη Συρία και το Ιράκ. Κύριε Μιγκαρέλη, σας καλωσορίζω. Θα μας ενημερώσετε τώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στην ε, Συρία και το Ιράκ. Ο κύριος Στάφαντε Μιστούρα, ειδικός ε, απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, προωθεί τοπικές ανακοχές ή καταπαύσεις πυρός, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ζώνες παγώματος προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό χρόνο που χρειάζεται η διεθνής κοινότητα για μια πολιτική λύση του, τη σύγκρουση στη Συρία. Η πρώτη ανακοχή θα μπορούσε να ξεκινήσει από το Αλέπο, το Χαλέπι, Πόλοι που ελέγχουν ε, η αντιπολίτευση και οι επαναστατικές δυνάμεις ε, και βρίσκεται υπό την πολιορκία των δυνάμεων του καθεστώτος της Συρίας. Ωστόσο υπάρχουν ε, φόβοι ότι το καθεστώς μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ανακοχές αυτές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία προκειμένου να ανακτηθεί ο έλεγχος στη Συρία. Για το Ιράκ υπάρχουν προσπάθειες για πολιτική σταθεροποίηση στη χώρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά και η τοπική περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν έχουν συμφωνήσει στα θέματα του προπολογισμού στις πληρωμές και τις εξαγωγές πετρελαίου. Μεγάλη πρόοδος προς ε, ε, εθνική φιλετική θρησκευτική ενότητα και δυνατότητα για το Ιράκ να αντιμετωπίσει το κίνδυνο του ISIS. Έχουμε λοιπόν το αίτημα του Οκτωβρίου προς μια περιφερειακή, συνολική περιφερειακή ε, πολιτική έναντι του κινδύνου για τη Συρία από το ISIS, από το Ισλαμικό κράτος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι δράσεις αναλογίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εν ώψη των συζητήσεων του Δεκεμβρίου για μια ευρωπαϊκή συνολική πολιτική και στρατηγική και θέλουμε να ακούσουμε τις θέσεις για τις τελευταίες εξελίξεις Συρία και το Ιράκ για τις προοπτικές σταθερότητας και ασφάλειας στη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή και θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι γίναμε μάρτυρες αυτό το Σαββατοκύριακο φρικιαστικών και αποτρόπιων πράξεων εις βάρος τόσο Αμερικανών υπηκών όσο και Σύρων στρατιωτών. Ο κίνδυνος λοιπόν από την ίσης ε, εξακολουθεί να υφίσταται στην περιοχή το Συμβούλιο, οπότε αντιλαμβανόμεθα σήμερα δεν υιοθέτησε συμπεράσματα ούτε για τη Συρία ούτε για το Ιράκ. Τώρα σας δίνω το λόγο, για 15 περίπου λεπτά μπορείτε να κάνετε την εισήγηση σας και μετά μπορούμε να συζητήσουμε με τους παρόντες συναδέλφους μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου προσφέρετε την ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων με τους ε, κυρίες και κυρίους βουλευτές για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την μάστιγα αυτή που έχει εγκύψει στη Μέση Ανατολή. Έχουμε να κάνουμε με μια δράκα βαρβάρων, πράξη αποτρόπες που των οποίων γίναμε μάρτυρε αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω πείθουν ότι η διεθνή κοινότητα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του συγκρατήσουμε. Πάνω από όλα αυτό σημαίνει με στρατιωτικά μέσα να εμποδίσουμε την προέλασή του και την επέκταση των δυναμεών του, γιατί σήμερα ελέγχουν το 1 τρίτο του Ιράκ αυτοί οι άνθρωποι, 1 τέταρτο τη Συρία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε πρώτη φάση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρεμποδίσουμε την προέλασή τους, την επέκτασή τους. Αυτό σημαίνει στρατιωτική επέμβαση. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο σχηματίστηκε ο συνασπισμό υπό του Αμερικανού με του Αμερικανού, αλλά και με συμμετοχή 60 κρατών όπω γνωρίζετε. ένα συνασπισμό, μια συμμαχία που εδώ και μερικέ εβδομάδε προβαίνει σε βομβαρδισμού θέσεων του λεγόμενου Ισλαμικού κράτου στο Ιράκ και τη Συρία και έχει επιτύχει τι τελευταίε εβδομάδε να παρεμποδίσει την προέλασή του. Σε ορισμένε περιπτώσει του υποχρώνει σε υποχώρηση. Άρα μπορούμε υπ' αυτή την έννοια να θεωρήσουμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της δράσης αυτής του διεθνούς, του συνασπισμού είναι μάλλον θετικά. Πολλοί σημειώνουν, και από εσά πιστεύω αρκετοί βουλευτέ, ότι δεν θα πρέπει αυτός ο συνασπισμός να γίνει αντιληπτός ως συμμαχία ε, δυτικών κρατών υπό τους Αμερικανούς, αλλά ως συνασπισμός κρατών αραβικών, κρατών μουσουλμανικών, στα οποία προσφέρουν ε, τη συνδρομή του στα ευρωπαϊκά ή τα δυτικά κράτη γιατί δεν θα μπορούσαμε να υπηρετήσουμε τώρα τα συμφέροντα και τους στόχους του, στόχου του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους ε, παρά μόνο ακριβώς ε, αφήνοντα να καθεδρυκθεί η ιδέα ότι έχει ξεκινήσει μια νέα σταυροφορία ει βάρο των Αράβων και Μουσουλμάνων. Τώρα λοιπόν αραβικά κράτη, μουσουλμανικά κράτη τα οποία στόχο έχουν να παρεμποδίσουν την προέλαση αυτών των βαρβάρων προχωρούν με την υποστήριξη των δυτικών κρατών. Φυσικά χωρίς την αμερικανική υποστήριξη θα ήταν ε, φαινάκι το να πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρεμποδίσουμε τις δυνάμεις αυτού του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, αλλά τώρα με την παρέμβαση και των Αμερικανών έχουμε πολύ θετικά μηνύματα. Οι ειδικοί στα στρατιωτικά, γιατί εγώ δεν είμαι, λένε ότι δεν αρκεί ο, η, ε, μια σειρά από βομβαρδισμού από αέρος, θα χρειαστεί η ανάπτυξη και επιγείων στρατευμάτων. Στο Ιράκ δηλαδή ένας νέος, νέο διαμορφωμένος στρατός Ιρακινός, αυτό είναι σαφές, για δε τη Συρία ακόμα είμαστε σε αναζήτηση αυτών των στρατευμάτων. Στο Ιράκ όμως οι Ιρακινοί με υποστήριξη κάποιων άλλων αρχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις ε, ταξιαρχίες και τις πολιτοφυλακές των ΣΥΙΤΟΝ που είχε αρχικά εγκαθιδρύσει ο Πρωθυπουργός Αλμαλική και τους μετατρέπουν σε Ιρακινό στρατό. Αλλά για να γίνει ένας πραγματικός στρατός αυτός του Ιράκ ε, χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά για να μπορέσει δηλαδή να αποκρούσει το, ε, το Ιζιλί Ίσης. Άρα λοιπόν υπάρχει στρατική παρέμβαση που είναι απαραίτητη, ε, είναι όρος οκτωνού κάμεφα αλλά όχι επαρκής. Χρειάζεται μια δράση αντιτρομοκρατική και μια σε διεθνές επίπεδο δράση. Για την καταπολέμηση του ΙΖΙΣ, αυτό που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ' όλα να επιδιώξουμε τη θέσπιση, την καθίδρυση μιας ε, στρατηγικής κατά των ε, λεγόμενων foreign fighters, των αλλοδαπών μαχητών, των ξένων μαχητών, αυτών που από τις χώρες μας φεύγουν για να πάνε στη Συρία και το Ιράκ, που αναλαμβάνουν, που λαμβάνουν τα όπλα δηλαδή στην ομάδα του ΙΣΙΣ και πρέπει να συνεργαστούμε στενά με την Τουρκία γιατί επί της ουσίας περνούν από τουρκικό έδαφος αυτοί οι μαχητές για να πριν φτάσουν στη Συρία και το Ιράκ. Έχουν μια σειρά επαφών με τις αρχές της Τουρκίας για να μπορέσουμε να ε, παρεμποδίσουμε να θέσουμε ε, μια τροχοπέδη στην άφηξη και διέλευση αυτών των μαχητών από τα ευρωπαϊκά κράτη. Χρειάζεται δράση και στον έλεγχο της τρομοκρατίας και στον έλεγχο των συνόρων. Στον έλεγχο των συνόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβεί σε επαφές με τις αρχές της Τουρκίας για να αναλάβουν δράση κυρίως όσον αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια της Τουρκίας και με τον τρόπο αυτό να επιβληθεί ένας ε, φραγμός, μια διαχωριστική γραμμή που δεν θα επιτρέπει την απροσκόπτη μετάβαση από την Τουρκία στη Συρία και του Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο και ίσως το μεγαλύτερο αγώνα είναι να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του κακού. Αυτό δηλαδή που επέτρεψε στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος να αναπτυχθεί και αυτό σημαίνει μια σειρά δράσεων στη Συρία και το Ιράκ. Για το Ιράκ μπορώ να σας το συνοψίσω σε λίγες ε, λέξεις. Πρέπει ο νέος Πρωθυπουργό Αλαμπάντη να πισθεί να προχωρήσει σε μια πολιτική ανοιχτή στην οποία θα, από την οποία δεν θα αποκλείονται ούτε οι Σουνίτες ούτε οι Κούρδοι μέσα στο Ιράκ και μια πολιτική η οποία θα εξασφαλίσει την ε, δίκαιη κατανομή του πλούτου στη χώρα προς δηλαδή και των Σουνιτών και των Κούρδων γιατί όπως γνωρίζουμε Εάν μεγάλο μέρος των Σουνιτών του Ιράκ ε, προσχώρησε στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, αυτό οφείλεται στην ε, πολιτική υπέρ του δόγματος των Σιητών, στην ε, διχοτομική πολιτική του προηγούμενου Πρωθυπουργού Αλμαλική που προσπαθούσε να προωθήσει τα συμφέροντα της Σιητικής κοινότητας, που οδήγησε έτσι σε μεγάλη απογοήτευση και στην των Σουνιτών και έτσι τους, έκανε, τους κατέστησε συμμάχους του Ισλαμικού κράτου, όπω ονομάζεται. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο νέο Πρωθυπουργό και να επιτρέψει τη συμμετοχή των Σουνιτών στην ε, άσκηση τη εξουσία, στα όργανα τη εξουσία και επίση να επιλύσει μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν που χρονίζουν και που ο Πρωθυπουργό Αλμαλική, ο προηγούμενο Πρωθυπουργό, είχε αφήσει να βαλτώσουν ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει πρώτον μεταφορά μέρου του Ομοσπονδιακού Προπολογισμού στι αρχέ του Κουρδιστάν Κουρδιστάν, προς τις αρχές του Κουρδιστάν. Δεύτερον, το ζήτημα των υδρογονανθράκων που είναι υποσυζήτηση για χρόνια τώρα, αλλά που δεν έχει οδηγήσει σε καταληκτική απόφαση. Είναι τρίτον, η διαπραγμάτευση για τις αμφιλεγόμενες ονομαζόμενες περιοχές, τις περιοχές του Κυρκούκ βασικά, αυτές που διεκδικούν τόσο το Κουρδιστάν όσο και το Ομοσπονδιακό κράτος του Ιράκ. Είναι πολύ σημαντικό ως εκ τούτου ο νέος Πρωθυπουργός να επιδείξει βούληση να αποδείξει βούληση που στέλνει την ε, λύση για να μπορούν Σουνίτες και Σιήτες και Κούρδοι να συμβιώνουν ομαλά και ειρηνικά στο Ιράκ. Ιδάλλως, ο κίνδυνος ε, είναι πολύ μεγάλος ότι θα γίνει στο μέλλον. Θα υπάρχει καν κράτος του Ιράκ, ε, γιατί είναι τόσο πολύ ευάλωτο το κράτος τώρα, είναι τόσο ασταθείς οι ρίζες του, που θα μπορούσαμε ακόμα και να δούμε κατάρρευσή του σε μικρότερα κράτη, διάλυσή του δηλαδή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ότι μπορείτε να διανοηθείτε. Η μετάβαση λοιπόν στην οικονομική και πολιτική μεταμόρφωση μέσα από μια συμμαχία συνεργασία που παράψαμε το Ιράκ ε, πριν από δύο χρόνια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέσα από αυτό θα το βοηθήσουμε. Είναι μια συμφωνία διαλόγου που θα μα επιτρέψει να προσφέρουμε υποστήριξη, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την καλή διακυβέρνηση, το κράτο δικαίου, για την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και των επενδύσεων όπω θα θέλαμε και επίση τομέα τη ενέργεια. Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε δραστηριότητε συνεργασία και συνεχή διάλογο με τις αρχές του Ιράκ. Αυτά ο ολίγης τα όσα προσπαθούμε να κάνουμε σε σχέση με τις αρχές του Ιράκ. Επίσης προσπαθούμε να τους πείσουμε να επιδείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και δράση ως προς τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπιστέντες που βρίσκονται μέσα στη χώρα. Ξέρω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι οι εκτοπιστέντες μαζί με τους πρόσφυγες που έχουν έρθει από τη Συρία στο Ιράκ. Μέχρι τώρα όμως οι αρχές της Βαγδάτης φαίνεται να μην μεριμνούν ιδιαίτερα για την μοίρα αυτών των ταλέπορων αντίθετα από ό,τι κάνουν οι κουρδικέ αρχές στο Ερβίλ που έχουν κινητοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσουμε στους Ιρακινού ότι οι εσωτερικά εκτοπιστέτε, όπως και οι πρόσφυγες είναι δική του δουλειά. Είναι δουλειά του κράτους του Ιράκ και πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών ώστε αυτοί οι δυστυχεί να μπορέσουν να ε, περάσουν το χειμώνα ω το δυνατόν πιο ανώδυνα. Για από τη Συρία τώρα η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη γιατί εξακολουθούμε να θεωρούμε πως δεν μπορεί να είναι εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση το καθεστώς του Ασάντ. Τι μας μένει, μας μένει μια λεγόμενη μετριοπαθής αντιπολίτευση την οποία πρέπει να βοηθήσουμε να εδρεωθεί πολιτικά αλλά και να ενισχυθεί στρατιωτικά. Ξέρουμε όμως από την άλλη, και δεν νομίζω ότι προσβάλλω κανέναν λέγοντας το δυνατά, ότι είναι μάλλον αδύναμη αυτή η μετριοπαθής αντιπολίτευση, είναι κατακαιρματισμένη, δεν μπορεί να σχηματίσει ενιαία πολιτική πλατφόρμα, στρατιωτικά δε η γραμμή της ε, διοίκησης φαίνεται ότι είναι πολύ ελλειπής. Ε, άρα λοιπόν άλλο να λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να τρέφουμε και ψευδεστήσεις, ίσως θα πρέπει να αναστήσουμε άλλες διεξόδους. Άλλες διέξοδοι λοιπόν τι θα ήταν ο κύριος Στάφαν ο ειδικό ε, εκπρόσωπος έχει διερευνήσει κάποιες λύσεις. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, προσπαθεί να πείσει το καθεστώς του Ασάντ να, σεβαστεί τις τοπικές ανακοχές και μάλιστα και μια, ένα πάγωμα των εχθροπραξιών περί την ε, πόλη του Χαλεπίου, πράγμα το οποίο θα μπορέσει να απαλύνει τα δεινά των πολιτών, των άμαχων που ζουν εκεί εδώ και 3,5 χρόνια μέσα σε πολύ δεινές συνθήκες ε, και μπορεί ταυτόχρονα να αναπτύξει αυτό και ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αμοιβαία συνεννόησης ενδεχομένως συν το χρόνο. Και έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία πολιτικών διαπραγματεύσεων και συνομιλιών μετά την αποτυχία του δεύτερου γύρου της Γενέβης πριν από ένα χρόνο και. Τώρα εδώ πρέπει να διαρωτηθούμε, αλλά βέβαια εγώ δεν μπορώ να δώσω από αυτή τη θέση απάντηση, γιατί μόνο υπάλληλο είμαι, δεν έχω τέτοια δουλειά, εάν θα πρέπει να επιμένουμε ως προς τις ε, προϋποθέσεις όπως την αποχώρηση από την εξουσία του Ασάντ, από την πρώτη στιγμή της μεταβατικής περίοδου, εάν θα πρέπει να επιδιώκουμε να κάτσουν οι άπαντες γύρω από την Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, ε, επί παραδείγματι λαμβανωμένου υπόψη ότι ο Ασάντ έχει μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία μέχρι τώρα με την υποστήριξη των Ρώσων και του Ιράν, άρα ίσως και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Μια σειρά λοιπόν από ερωτηματικά που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, να τα συζητήσουμε και βέβαια σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση, διότι εάν δεν αναζωογονηθεί η διαδικασία για πολιτικές συνομιλίες, είναι αδιανόητο στους επόμενους μήνες να περιμένουμε ότι θα σταματήσουν οι σφαγές, οι εκατόμβες αυτές που εδώ και 3,5 χρόνια ε, βλέπουμε στη Συρία. Αυτό μπορούμε να προσπαθήσουμε στη Συρία. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να λησμονούμε τους γείτονες Λίβανος, η Ορδανία, χώρες οι οποίες έχουν αποδυναμωθεί ιδιαίτερα και βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση λόγω της κρίσης στη Συρία. Ο Λίβανος έχει ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, ε, διέρχεται μια πολύ σημαντική πολιτική κρίση. Προσπαθούμε να προσφέρουμε με ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και με αναπτυξιακή βοήθεια, υποστήριξη. Ενισχύουμε τις δυνατότητες τους για ενίσχυση των βασικών ε, δομών όπως εκπαίδευση και υγεία. Οι αρχέ της Ιορδανίας επίσης ε, θα έπρεπε να λάβουν όλοι μας την προσοχή και υποστήριξη. Αυτά εν ολίγης και μέσα σε 15 λεπτά κύριε Πρόεδρε όπως μπορέσα να συνοψίσω την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαγκαρέλη για την πληρέστατη αυτή παρουσίαση. Να δώσω το λόγο αρχικά από πλευρά ε, Έλκα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. κυρία Λίο Μαρή. Θα ήθελα να μας ε, πείτε αρχικά ποια είναι η εκτίμησή σας για τις παρεμβάσεις, είτε αυτές είναι προφανείς είτε συγκεκαλυμμένες, του Ιράν και, και μια σειρά άλλων χωρών του Αραβικού κόλπου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ρίτσαρτ Χάουιτ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Μιγαρέλη που βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Να σας δώσω δύο λεπτά να βάλετε ακουστικά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ενημέρωση. Το πρώτο ερώτημα είναι, Ακούσαμε το προσοχή σε την ανάλυση σας. Θα ήθελα να είστε λίγο πιο συγκεκριμένο για τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το συνασπισμό, σε αυτή τη συμμαχία. Τι, πώς συνεισφέρουμε εμείς σε αυτό το συνασπισμό. Ποια είναι η δική μας συμβολή. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ευρία βάση για αυτό το συνασπισμό, αλλά να ξέρουμε ότι κατά πόσο απλώς ε, μιλάμε για στήριξη ή κατά πόσο το εννοούμε πραγματικά. Και υπάρχουν και ιδιαιτερότητε σε ό,τι αφορά τον ε, ρόλο επιμέρους κρατών μελών για τυχόν ε, συνδρομή στον τομέα της προστασίας που ενδεχομένως να ε, παράσχουμε. Αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά στην παρουσίασή σας, είναι η αποτελεσματικότητα των δυνάμεων επιτόπου. Είναι θεμελιώδες στοιχείο της υπόθεσης. Και μετά, Ποια είναι η δική σας εκτίμησή σα ε, για ε, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, για την συνδρομή ως προς την ασφάλεια σε αυτές τις δυνάμεις. Μιλήσατε μετά για συμφωνία μεταξύ των αρχών της Βαγδάτης και αρχών στο Ερμπίλ για τα έσοδα από το πετρέλαιο. Πριν από μερικές εβδομάδες, πολλά υπόθηκαν για κάποιες ενέργειες ε, του Κουρδιστάν και στο βόρειο τμήμα του Ιράκ και κατά πόσο πρόκειται για αποσχιστικές τάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο το θεωρείτε ε, κρίσιμη σημασία σε όλα αυτά τα στοιχεία για την ε, κατάσταση ό,τι αφορά το Ιράκ και αν υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις στο βορρά. Τη δική σας ανάλυση θα ήθελα. Και τέλος, πολλά υπόθηκαν στην Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο για το ρόλο της Τουρκίας και γιατί η Τουρκία δεν συνεργάζεται μαζί μας ε, για τον ISIS. Θίξατε το ζήτημα των ε, foreign fighters ε, και της αντιτρομοκρατικής συνεργασίας, αλλά θα ήθελα να είστε πιο συγκεκριμένος αν μπορείτε για το πώς κατά πόσο μάλλον η Τουρκία διαδραματίζει σημαντικό και αξιόπιστο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, Κάποιοι μίλησαν για τον αγκαίο κακό της συνεργασίας με τον Ασάντ, δεδομένη της απειλής του ISIS. Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά θεωρεί ότι ο Ασάντ είναι εν δυνάμει ε, εγκληματίας πολέμου και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ακριβώς αυτό το στοιχείο. Πρέπει να δούμε πάντα πώς ε, μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Κάποιοι βεβαίως διαφωνούν και θα ήθελα να ε, μιλήσετε επισήμως, να μας δώσετε τη θέση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ κύριε Χάουετ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ντεμεσμάκερ. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μεγαρέλη για την ε, ενημέρωση. Βέβαια μέσα στα 15 λεπτά είναι δύσκολο κάποιος ε, να αναλύσει και να παρουσιάσει μια τόσο ε, περίπλοκη σύγκρουση. Βλέπουμε ότι είναι πολύ ε, πολύπλοκα τα πράγματα λοιπόν και το καταλαβαίνουμε αυτό κάθε μέρα. Μια συνολική στρατηγική λοιπόν είναι απαραίτητη εδώ και τώρα. Οι αεροπορικές επιδρομές ε, του συνασπισμού της συμμαχίας αυτής επικεντρώνονται σε στόχους ε, του ISIS στην περιοχή του Κουρδιστάν. Ο ελεύθερος Ιρακός στρατός ζητά ε, να πληγούν στόχοι και του καθεστώτος Ασάντ. Για κανέναν δεν είναι σαφές. Ναι, λέτε ψάχνουμε εταίρους, συμμάχους στη Συρία. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πόσοι από αυτούς τους ε, αρχικούς ε, αντιστασιακούς ε, ε, στη Συρία συνεχίζουν να αγωνίζονται με, κατά ποιου αγωνίζονται μεταξύ του ενάντια στον Ασάντ, ενάντια στον ε, Ίσης μήπως και αυτοί διαπράττουν εγκλήματα πολέμου. Κανένας δεν το γνωρίζει αυτό αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλά ερωτήματα προς αυτό. Πριν από μερικέ ημέρες ή εβδομάδε ακούσαμε και του ίδιου του Κούρδους εδώ και εκείνοι ζητούν ε, ενδυνάμωση, στήριξη, ζητούν όπλα. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο και σε, σχέση με τις, ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία, αλλά ποια είναι η δική σας γνώμη προς αυτό. Και κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένως για για το κατά πόσο θα συμμαχίσουμε ή όχι με το καθεστώς Ασάντ είπατε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Αλλά εσείς προσωπικά τι θεωρείτε, ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος ε, ορισμένων χωρών για να εξευρεθεί λύση. Υπάρχει πραγματικά τέτοια συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ε, πόσο εκτιμάτε εσείς τον κίνδυνο ε, μετάγγισης του ζητήματος ε, και στο Κάιρο, στην Αίγυπτο. και τι κάνουμε ως προς τη χρηματοδότηση του ISIS, του Ισλαμιστικού κράτους. Γιατί κατάφεραν πολύ γρήγορα να σημειώσουν επιτυχίες και να θεμελιώσουν τη θέση τους και αυτό χάρη στη δυνατότητά τους να λάβουν, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και μέσω ε, του πετρελαίου τι κάνουμε εμείς για να αποκόψουμε αυτές τις, ε, τις πηγές χρηματοδότησης ε, της οργάνωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Ντεμεσμάκερ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νέιτς. Συνάδελφοι, έχουμε άλλα 35-40 λεπτά το πολύ, οπότε τρίλεπες τοποθετήσεις παρακαλώ, γιατί στον κατάλογο ομιλητών έχω ήδη 11. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαγκαρίνη για την παρουσίαση. Θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη του σε ό,τι αφορά την ανάλυση ε, κάποιων αντιπολιτευμένων στο Ιράν που διατείνονται ότι σήμερα το καθεστώς Αστάντ έχει παραδοθεί απολύτως στο Ιράν βρίσκεται υπό την απόλυτη επιρροή λοιπόν του Ιράν σε στρατιωτικό, οικονομικό, στρατηγικό επίπεδο. Δεν υπάρχει πλέον καθεστώς. Και, ότι, και αυτοί οι αντιπολιτευόμενοι προσθέτουν και ένα αρκετά αρνητικό στοιχείο. Αναφέρουν ότι κάποιοι, υποπτεύονται τουλάχιστον, ότι κάποιοι δυτικοί δεν το βλέπουν και με τόσο κακό μάτι αυτό που συμβαίνει. δηλαδή, ότι μπορεί να είναι και θετικό το να το αναλάβει πλήρως το Ιράν το ζήτημα. Ε, εγώ δεν ξέρω κατά πόσο να δεχθούμε αυτή την, ε, αυτόν τον ισχυρισμό. Εσείς τι εκτιμάτε. Υπάρχει πράγμα τέτοια επιρροή του Ιράν στο καθεστώς Ασάντ. Αυτό ισχύει και για ε, τη Συρία και σε ό,τι αφορά το, τη Χεσβολά. Εσείς τι ακριβώς πιστεύετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μέτς. Λοχ Βιλέρ Βάρβελα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλ για την ενημέρωση. Στην ομάδα των Πρασίνων την τελευταία εβδομάδα κάναμε μια ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολευτών στη Συρία και με μετροπαθείς δυνάμεις και καταγράψαμε ότι στη δική σας αντίληψη ο αγώνας κατά του Ισλαμικού κράτους ε, επικεντρώνεται ε, στο Ιράκ αλλά ε, ε, αλλά δεν αναφέρονται ιδιαίτερα τα ε, εγκλήματα που διαπράττονται στη Συρία και από το καθεστώς Άσαντ και ε, υπήρχαν και πολύ σωστά και καλά επιχειρήματα. Πώς εσείς λοιπόν διασφαλίζεται ότι ακούγονται οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών ε, στην δική σας στρατηγική, πώς εντάσσονται οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών στη δική στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Άννα Γκόμες παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you for being, uh, for what you told us. Ευχαριστώ κύριε Μιγκαρέλη για όσα μας είπατε. Πρώτα απ' όλα να σας πω πόσο θλιβερό είναι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση και τα κράτη-μέλη δεν είναι ακόμα σε θέση να διοργανώσουν μέσα σε ένα πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής μια συντονισμένη δράση και να λειτουργήσουμε σωστά με τους εταίρους μας, είτε με τους ε, Αμερικανούς, τον ΙΠΑ, είτε με Άραβες εταίρους. Και πραγματικά αυτό δείχνει πόσο εκτρή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη και θα έπρεπε να ντρέπονται οι κυβερνήσεις μας. Εγώ τουλάχιστον ντρέπομαι. Θα ήθελα να ζητήσω να υποστηριχθεί η δράση του κυρίου Ντεμίστουρα που πραγματικά είναι πολύ έμπειρος, πεπειραμένος ε, σε σχέση με αυτή την περιοχή και έχουμε περισσότερους ε, ικανούς ε, από ό,τι είχαμε πριν από δύο χρόνια. Όταν πήγα στα σύνορα της Γκαζιαντέπ στην Τουρκία με τα Συριακά σύνορα κοντά, στο Αλέπο κοντά και είχαμε την ανακυκλούμενη, ας το πω έτσι, την, ε, το εξανακυκλώσεως σύστημα, το οποίο ήταν ικτρό. Πραγματικά θλιβερό να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους επιμελητιακή υποστήριξη ή πολιτική συνδρομή όσον αφορά ε, την προσπάθεια που γινόταν τώρα με την προσπάθεια του κυρίου Ντεμίστουρα σε σχέση με αυτό το θέμα του Αλέπο. Μετά για το Ιράκ. Πραγματικά υποστηρίζω όλα όσα είπατε σε σχέση με τα όσα πρέπει να γίνουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά και πάλι, τι κάνει ο πρέσβης μας συνεχίζει να περιορίζεται στη Βαγδάτη και στην, ε, στα κτίρια της Βρετανικής ε, Πρεσβείας και δεν μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή και να συζητήσει με τους ε, KRG και είναι η ίδια κατάσταση. Δεν φταίτε εσείς βέβαια, αλλά και πάλι είναι ολέθρια η κατάσταση και ελπίζω ότι μπορείτε να διαβιβάσετε στη νέα το εκπρόσωπο πραγματικά ότι αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, ταχύτατα. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι αποτελεσματική και δεν θα καταφέρει τίποτα. Αναφέρθηκε το ζήτημα του Ιράν και το Ιράν είναι εμπλεκόμενη δύναμη σε αυτή την περιοχή και θα μπορούσε να έχει κοινό συμφέρον στο να μπορέσει να καθοριστεί, να αντιμετωπιστεί το θέμα των ε, Σουνιτών, ε, των Σαλαφιστών, εξτρεμιστών ε, στις ακραίες δράσεις τους. Και πάλι έχει γίνει κάτι, έχει υπάρξει κάποια επαφή, ανιχνευτική επαφή με το Ιράν ώστε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πώς θα μπορούσε να εμπλακεί το Ιράν ώστε να δράσει σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν με τον Ασάντ και τι θα μπορούσε να συμβεί. Και τέλος, όσον αφορά και τον ελέφαντα στην αίθουσα που είναι πολύ πιο κοντά σε μας, η Λιβύη και βλέπουμε ότι και εκεί πάλι δρούν οι ακραίοι Ισλαμιστές ε, με αποκεφαλισμούς ε, και είναι πάλι μια ικτρή αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανέναν δεν μπορούμε να, ε, σε κανέναν δεν μπορούμε να αποδώσουμε το φταίξιμο. Δικό μας είναι. Τι κάνουμε. Κάνουμε όσο, όσα μπορούμε και πάλι εδώ σε σχέση με την αποστολή Ηνωμένων Εθνών πρέπει να υποστηρίξουμε τη δράση αυτή όμως η κατάσταση είναι ικτρή Ποιος είναι ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας, ε, της Αιγύπτου, του Κατάρ στη Λιβύη και τι κάνουμε. Απλά σταυρώνουμε τα χέρια και προσπαθούμε να σώσουμε κάποιους ε, μονομένα άτομα ενώ βυθίζεται, καταποντίζεται ε, το σκάφος στη Λιβύη και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να μην αναφέρω και την ικτρή κατάσταση των Λιβύων των ιδίων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιούρεκ, παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ. Ήθελα να θέσω ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την ε, κατάσταση της χριστιανικής ε, κοινότητας. Γιατί ενημέρωση λαμβάνουμε μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να Παρακολουθούμε στενά ε, την κατάσταση ότι αφορά τη χριστιανική κοινότητα γιατί ε, πρέπει να δείξουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Επομένως, θα θέλαμε κάποιες ε, πληροφορίες και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να την προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιούρεκ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Στερεβίτσιους. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μιγκαρέλη, σας ευχαριστώ πραγματικά για την ενημέρωσή σας, για τα ζητήματα που είμαι σίγουρος ότι εδώ και χρόνια απασχολούν ε, την υπηρεσία σας και κατανοούμε βεβαίως και τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Έχω δύο ερωτήματα να σας θέσω. Πρώτον, οι φλόγες γύρω από μια χώρα που δεν αναφέρθηκε επαρκώς ε, είναι γύρω από το Ισραήλ και η εισβολή ξένων μαχητών, βρώμικης χρηματοδότησης από γειτονικέ χώρες, από το Λίβανο, την Ιορδανία και σε μεγάλο βαθμό και από την Αίγυπτο, ε, πώς ε, άλλαξαν όλα αυτά τα στοιχεία τον ε, διάλογο για θέματα ασφάλειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατική χώρα στην περιοχή. Έχει δικά του συμφέροντα όσον αφορά την ασφάλεια και σε ποιο βαθμό θα μπορούσατε να μας σχολιάσετε ε, τον διάλογο υπό το φως της κατάστασης ασφάλειας που έχει αλλάξει στην περιοχή. Οι χώρες του κόλπου έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι χώρες αυτές είναι πρόθυμες να συνεργαστούν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση προκλήσεων, ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Υπάρχουν απτές ανταλλαγές πληροφοριών που αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η συνεργασία για να βελτιωθεί η κατάσταση. Βλέπετε τουλάχιστον να, ε, ή έχετε εσείς μάλλον από τη δική σας πλευρά ε, πολιτικό ενδιαφέρον για να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σεμπάλους έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται. Βελτιώθηκε η βοήθεια αυτή, βελτιώθηκαν τα πράγματα, φτάνει πράγματι στον προορισμό της. η βοήθεια αυτή θα έπρεπε να καταλήγει σε ένα βαθμό και στις γειτονικές ε, χώρες. Επίσης, ως προληπτικά μέτρα, αν θέλουμε να αποδυναμώσουμε το Ισλαμικό κράτος, θα πρέπει να στεγνώσουμε, να ε, στραγγαλίσουμε τις ε, πηγές του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχουν χώρες που τροφοδοτούν το Ισλαμικό κράτος. Υπάρχουν οικογένειες, για παράδειγμα, που με τα παιδιά τους πηγαίνουν στο Ιράκ και στη Συρία για να στρατολογηθούν ε, νέοι άνθρωποι, τα παιδιά τους, οι ίδιοι, στο Ισλαμικό κράτος. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποτρέψουμε... Ε, να δημιουργείται η αντίληψη σε νέους ανθρώπους ότι το Ισλαμικό κράτος είναι το μέλλον τους. Και επίσης μιλήσατε για την Εθνική ε, Συμμαχία ε, της Συρίας. Εξακολουθεί να είναι ο επίσημος συνομιλητής μας παρά το γεγονός ε, του ότι έχουν εμφανιστεί, παρά το γεγονός ότι έχουν εμφανιστεί συγκεκριμένα προβλήματα. Επίσης, είπατε ότι έχουν ε, κινητοποιηθεί τα πράγματα στην, στο Ιράκ. Περιμέναμε πολύ καιρό γι' αυτό, αλλά θεωρείτε ότι το Ιράκ θα αντέξει ή μήπως στο μέλλον θα αποκτήσουμε, θα έχουμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον με τρία διαφορετικά κράτη. Ευχαριστώ κύριε Σομπάλος και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάν, συνάδελφο κύριο Κάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω και για τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με το Ιράκ αλλά και το Ισλαμικό κράτος. Σε σχέση με το Ιράκ, είπατε ότι ε, οι ΙΠΑ εκπαιδεύουν τον Ιρακινό στρατό. Αυτό δεν συνέβαινε και προτού χορηγηθούν 25 ε, δισεκατομμύρια για την αγορά όπλων. Γιατί πιστεύετε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα, θα, θα στεφτούν με περισσότερη επιτυχία. Επίσης, θα γίνει δημοψήφισμα στο Ιράκ από τους Κούρδους. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτού του δημοψηφίσματος ε, στο Ιράκ όσον αφορά το Ισλαμικό κράτος. Ε, χαιρετίζω βεβαίως τη συμμετοχή των αραβικών κρατών στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους και είναι σημαντικό να φανεί ότι βρίσκονται εκείνα τα κράτη, τα αραβικά, στην εμπροσθοφυλακή. Αλλά όσον αφορά τον, <coughs> τον Άζατ, πιστεύω ότι το Ισλαμικό κράτος συνδέεται με τον Άσαντ Ανησυχώ και για τους 3.000 ε, υπηκόους Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, στρατολογήθηκαν στο Ισλαμικό κράτος και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ένα, ένα από τα social media που χρησιμοποιούνται Ποια είναι τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε τη στρατολόγηση νέων ανθρώπων από την Ευρώπη και τι είδους συμβουλές και βοήθεια δίνουμε στους γονείς, δεδομένου ότι και οι γονείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Έχετε κάποια στρατηγική, έχετε επεξεργαστεί κάποια τακτική, μάλλον για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Και ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Νάρτ. Ευχαριστώ πολύ. Η Σύρια και το Ιράκ είχαν τις πιο προηγμένες κοινωνίες με έναν πολιτισμό υποδειγματικό θα έλεγα για τη Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή έχουν μετατραπεί σε κέντρα αδιαλαξίας και σε σχέση με τους, τις διάφορες θρησκείες, αλεβίτες, δρούσους που υπήρχε ανοχή σήμερα υπάρχει απογοήτευση και είναι απόγνωση που επικρατεί και συνεχίζουμε δυστυχώς. Είναι, υπάρχει τυφλότητα που συνεχίζεται σε σχέση με αυτήν την κατάσταση και στο Ιράκ και στη Συρία. Είπατε υπάρχει μια νέα κυβέρνηση στο Ιράκ που λέει κάτι το οποίο είναι αληθινό. Αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τους πρόσφυγες. Και είπε ότι είτε είναι Σουνίτες είτε είναι οποιοδήποτε οι μετανάστες όμως οι πρόσφυγες με συγχωρείτε για τους Σιήτες με την ε, νέα κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει τίποτα είναι αδιάλακτη και είναι μεροληπτική όπως ε, με την κυβέρνηση του Μαλίκη και με μια τέτοια μεροληπτική κυβέρνηση πολύ λίγα μπορούν να γίνουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε αυτή η κυβέρνηση που παίρνει τεράστια βοήθεια από εμάς να μπορέσει να δράσει ως κυβέρνηση του Ιράν και όχι ως μεροληπτική κυβέρνηση των δικών της ανθρώπων, των Σιητών. Δεύτερον, στην ε, Συρία θα πρέπει να μην καταστραφεί η ελπίδα σε σχέση με αυτή την αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη όσον αφορά την ε, αντίσταση στη Συρία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία προοπτική για μια άλλη εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική λύση για τον ε, έναντι του Ασάτ που είναι ένα, μια εγκληματική κυβέρνηση. Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάτι για να προαχθεί μια πραγματική εναλλακτική λύση που δεν θα είναι η Ισλαμική λύση, η μόνη λύση με μια, σε σχέση με μια προηγμένη κοινωνία όπως ήταν η κοινωνία της Συρίας. Μετά τέλος έχουμε την ε, Τουρκία που είναι κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή και είτε μας αρέσει είτε όχι και το Ιράν ε, είναι κυρίαρχη δύναμη και πρέπει να το δεχθούμε αυτό σε σχέση με τη Συρία. Ερώτηση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία και τι, ποιες συμφωνίες υπάρχουν ή ποιες δυνατότητες συμφωνιών υπάρχουν Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο και σύνθετο το θέμα. Υπάρχει μια αντιφατική κατάσταση. Επειδή υποστηρίζει το Ιράν το καθεστώς ε, του Ασάντ. Υποστηρίζει τη Χεσμολά που υποστηρίζει τον Ασάντ. Όμως ακόμα και έτσι το Ιράν είναι ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Τι κάνουμε με αυτούς λοιπόν. Ευχαριστώ. thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νάρτ. Νομίζω ότι κάναμε το γύρο όλων των συναδέλφων που ήθελα να μιλήσω. Θα παρακαλώ τώρα τον κύριο Μέγκαρελή να απαντήσει στις ερωτήσεις. Έχουμε άλλα 15 με 20 λεπτά στη θέση μας. Άρα θα έχετε αρκετό χρόνο, πιστεύω. Ήταν πολλέ ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τι ερωτήσει που ακούστηκαν. Ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα. Για την κυρία Αλιομαρή που μας ε, ρωτάει πώς συμπεριφέρεται το Ιράν ε, και οι χώρες του Περσικού. Για το Ιράν η κατάσταση είναι σχετικά απλή. Υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα τον Ασάτ και το καθεστώ του, για τη Συρία μιλάμε, και είναι αναμφίβολο ότι χωρίς την υποστήριξη του Ιράν δεν θα ήταν πια στην εξουσία στη Δαμασκό ο Ασάτ διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο επίσης όσον αφορά τη στρατιωτική ηγεσία, η αλυσίδα της ηγεσίας του στρατού, από ό,τι μας λένε οι στρατιωτικοί παρατηρητές, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Δαμασκό, απαρτίζεται από Πασδαχάν και φύλακε της επανάσταση του Ιράν. Άρα χωρίς την υποστήριξη του Ιράν και σε βαθμό συγκεκριμένο και χωρίς την υποστήριξη του Χεσμολάχ θα ήταν διαφορετική η συσχετισμή δυνάμεων στη Συρία. Άρα εδώ έχουν ξεκάθαρα επιλέξει ε, ποιον υποστηρίζουν οι Ιρανοί. Για τις χώρες του Περσικού. Η εικόνα είναι λιγότερο σαφής στη Συρία. Γιατί εάν σήμερα το Ισλαμικό κράτος και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες όπως το μέτωπο Αλνούστρα ε, βρίσκονται εκεί που βρίσκονται τώρα, αυτό οφείλεται ότι έλαβαν εξωτερική βοήθεια. Από πού ήρθε αυτή η βοήθεια? Είναι αρκετά πιθανόν πάντως μέρος της βοήθειας να προέρχεται από την Μέση Ανατολή. Είναι αρκετά πιθανόν. Και μάλιστα αυτό ίσως δεν προέρχεται απαραίτητα από τις εθνικές αρχές των εμπλεκομένων κρατών, αλλά είναι πολύ πιθανό ιδιωτικές πηγές, ε, ε, ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, charities, να έχουν προσφέρει ε, εξοπλισμό σε αυτούς που τώρα είναι μέσα στο Ισλαμικό κράτος ή στο μέτωπο Αλνούσρα. Είναι αρκετά πιθανόν. Ταυτόχρονα οι χώρες του Περσικού αισθάνονται αυτή τη στιγμή απειλούμενες από αυτόν τον εξτρεμισμό, τον σουνητικό εξτρεμισμό, γιατί ξέρουν ότι είναι και θύματα της Ντάσο, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, η ίσης, και άρα συμμετέχουν τώρα στον ε, διεθνή συνασπισμό για να βοηθήσουν ε, να εξολοθρευτεί το Ισλαμικό κράτος. Άρα, ναι μεν τώρα συμμετέχουν στην ε, συμμαχία αυτή, στο συνασπισμό αυτών διεθνή, αλλά είναι πολύ πιθανό να προσέφεραν παλαιότερα όπλα χωρίς να κοιτάνε πολύ προσεκτικά ποιος ήταν αυτός τον οποίο κατέληγα, κατέληγαν τα όπλα. Τώρα όμως αντιλαμβάνονται ότι το Ισλαμικό κράτος αποτελεί απειλή για τα ίδια, για τους ίδιους και έτσι συμμετέχουν στο διεθνή συνασπισμό για να βοηθήσουν να εξολοθρευτεί αυτό το, αυτή η οργάνωση. Ο ρόλος της Ένωσης, κύρια Χάουιτ, στο συνασπισμό. Ε, έχουμε αφενός με το ρόλο των κρατών μελών χωριστά και της Ένωσης αυτής καθευτής. Ως προς τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν 8, 8 κράτη-μέλη που είτε συμμετέχουν στα πλήγματα είτε προσφέρουν εξοπλισμό ε, οκτώ κράτη-μέλη επαναλαμβάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που μπορεί να προσφέρει είναι ε, η πολιτική υποστήριξη για να ενισχυθεί ο συνασπισμός. Πώς ταξιδεύουμε στα κράτη που βρισκόνται κοντά στη Συρία και το Ιράκ, στα αραβικά κράτη, στη Συρία, για να εξηγήσουμε πόσο ε, θα πρέπει να ενστερνιστούν αυτόν το συνασπισμό, πόσο αφορά τα ίδια κράτη ο συνασπισμός και θα πρέπει να συμμετάσχουν στον αγώνα. Ε, χωρίς τον οποίο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επεκταθεί το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος και το μέτωπο Αλνούσρα με πρώτους πληττόμενους αυτούς τους ίδιους, αυτά τα ίδια κράτη. Αυτό νομίζω, με αυτόν τον τρόπο μπορώ να συνοψίσω τον ρόλο της Ένωσης. Δηλαδή είναι πολιτικός ο δικός μας ρόλος. Προσπαθούμε να ε, ενισχύσουμε, να εδραιώσουμε τον συνασπισμό με τη δύναμη της πυθούς ε, στη συνεργασία με τους περιφερειακούς παράγοντες και χώρες περιφερειακές ε, να ενισχυθεί αυτός ο συνασπισμός, να γίνει πιο αραγής και ταυτόχρονα βέβαια να ενισχυθεί και η θέση των δικών μας κρατών. Συμφωνίες ε, του Ερμπίλ και Βαγδάτη και αν σημαίνουν ότι έχει σφραγιστεί για χρόνια πια το πεπρωμένο του Ιράκ και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διάλυσης. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να το ισχυριστώ επουδενή. Ξέρουμε ότι ο τελικός στόχος των Κούρδων είναι η ίδρυση ανεξάρτητου κράτους. Ο δικός μας ρόλος όμως είναι, ότι θα πρέπει να, είναι να τους υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να παραμείνει ενωμένο το Ιράκ, να διαφυλαχθεί η εθνική του κυριαρχία, η ακεραιότητά του ε, και να πείσουμε τους Κούρδους ότι μπορούν να έχουν μέσα σε ένα Ιρακινό κράτος μεγάλο βαθμό αυτονομίας. Ένα Ιρακινό κράτος το οποίο θα εξασφαλίζει την, ε, τον επιμερισμό του πλούτου μέσα σε ένα κράτο προ όφελο τόσο των Ιρακινών όσο και του κουρδικού λαού. Αν και ομολογώ ότι δεν είμαι βέβαιο ότι αυτό θα αρκέσει για να μείνει το Κουρδιστάν μέσα στου κόλπου του Ιράκ στην προσεχή 20 ετία. Πάντω, βράχει και μέσω πρόθεσμα, αυτό είναι ο αγώνα μα. Τουρκία. Ο ρόλος Τουρκίας ήταν αμφίσιμος για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εξελιχθεί. Ξέρουμε ότι πριν από δύο-τρία χρόνια ακόμη οι Τούρκοι άφηναν να περνούν ξένοι μαχητές από το έδαφος τους. Μετά διαπίστωσαν ότι αποτελεί για τους ίδιους απειλή το Ισλαμικό κράτος και έτσι τώρα συνεργάζονται μαζί μας και με τους υπόλοιπους στο συνασπισμό για καλύτερη προστασία των συνόρων και για τα καταπολέμηση των ροών αυτών των ξένων μαχητών. Με τον ίδιο τρόπο οι Τούρκοι συνεργάζονται μαζί μας τώρα και με κάποιους άλλους για να προσπαθήσουν ε, να διαβρώσουν τις πηγές χρηματοδότησης του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους και κυρίως μέσω του, ε, της καταπολέμησης του λάθρεμπορίου προϊόντων πετρελαϊκών από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτο. Άρα έχουν ένα σαφή ρόλο πλέον. Ο κύριο Δεσμέκερ μα λέει ότι πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια στου Κούρδου. Ναι, βεβαίω έχετε δίκιο, πρέπει να του βοηθήσουμε και στο Ιράκ. Πρώτα απ' όλα για το Ιράκ τώρα, οι Κούρδοι είναι εκείνοι που υποδέχονται το μεγαλύτερο κομμάτι των ε, εκτοπιστέντων και προσφύγων και το κάνουν με μεγάλη γενεοδορία. Το είδα και η σώμασιν σε επίσκεψή μου στο Ερμπίλ, όπου είδα πως η περιφερειακή κυβέρνηση κινητοποιείται για να προσφέρει κύρια βοηθεία σε αυτούς τους ε, ε, Δυστυχής, άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε για να αντιμετωπίσουν αυτό το ανθρωπιστικό πρόβλημα που έχουν μπροστά τους, αλλά επίσης και τους Κούρδους του, της Συρίας πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί ξέρετε ότι οι δυστυχείς κάτοικοι του Κομπάνη έχουν γνωρίσει ζωφερή μοίρα, πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και αυτούς τους Κούρδους της Συρίας όταν απειλούνται από σφαγές. Κούρδοι της Τουρκίας. Ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πιο περιπλοκή, γιατί το ΠΚΚ χαρακτηρίζεται ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρομοκρατική κόκκινημα. Έχουμε πάντως υποστηρίξει εντωμεταξύ τον διάλογο που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση Ερντογάν πριν από ένα διάστημα με τους Κούρδους. Βεβαίως και θέλουμε η αντιπαράθεση μεταξύ της εξουσίας της Άγκυρας και των Κούρδων να επιληθεί μέσω ενός εσωτερικού διαλόγου στην Τουρκία. Για την κυρία Νέιτς. Απάντησα στις ερωτήσεις σας αν το καθεστώς Ασάντ είναι στα χέρια των Ιρανών 100%. Σας απάντησα ήδη και άλλωστε αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα τα πράγματα θα σας επιβεβαιώσουν ότι χωρίς την υποστήριξη των Ιρανών δεν θα ήταν εκεί που είναι τώρα ο Ασάντ, δεν θα ήταν στην εξουσία ακόμα και πρέπει να δούμε όταν έρθει η στιγμή πώς θα επιτρέψουμε στους Ιρανούς να συμμετάσχουν στο μεγάλο διάλογο που θα πρέπει να γίνει για την επαύριον Ξέρω ότι τώρα δεν είναι η ώρα να γίνει αυτή η συζήτηση και θα επικεντρωθούμε κυρίως στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να δούμε και το θέμα αυτό και τη θέση των Ιρανών σε μια παγκόσμια διαπραγμάτευση, σε μια γενικότερη καλύτερη διαπραγμάτευση. Χωρίς τους Ρώσους το ίδιο θα συνέβαινε και παρά τις όποιε δυσκολίες ε, έχουμε σε σχέση με την Ουκρανία, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι Ρώσοι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη Συρία και ότι αν αύριο θέλουμε να ξαναδώσουμε όθηση σε έναν πολιτικό διάλογο και να του επιτρέψουμε και να καταλήξει μια επιτυχή ε, έκβαση, πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι Ρώσοι και να είναι μέρος της συνολικής λύσης. Η κυρία Λόχμπίλερ μας ρώτησε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, ε, φωνή της κοινωνίας των πολιτών Πώ μπορούμε να παρακολουθούμε τη λέει η κοινωνία των πολιτών. Κοιτάξτε, εμεί έχουμε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών και με την μετριοπαθή αντιπολίτευση τη Συρίας, χωρί αυτό να σημαίνει ότι αρκούν όλα αυτά, πάντα μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο, αλλά σα βεβαιώνω ότι έχουμε τη βούληση να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η κοινωνία των πολιτών και η μετριοπαθή ε, αντιπολίτευση να συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγική μα και να ωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την ανθρωπιστική και μη ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή τη ε, συνεργασία για την ανάπτυξη που προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει προ όφελο του πληθυσμού τη Συρία. Για την κυρία Γκόμε, μου θέσατε ερωτήσει που με φέρνουν σε αμηχανία και δεν ξέρω και τι να απαντήσω. Πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο, στο Βρετανικό στρατόπεδο, στο Ιράκ. Όντω, ναι. Έτσι είναι άλλες επιλογές, τι να σα πω, μπορεί και να υπάρχουν. Ελπίζω κάποια στιγμή να μελετηθούν πιο προσεκτικά και σχετικά σύντομα, να δούμε αν υπάρχουν άλλες επιλογές για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Φαντάζεστε βέβαια και εσεί ότι είναι πολιτικέ οι αποφάσει. Για το Ερμπίλ, αν χρειάζεται να στείλουμε κάποιον, ναι, ασφαλώ. Θα ήταν χρήσιμο τουλάχιστον μπορώ να πω. Προ το παρόν έχουμε τακτικέ επισκέψει των συναδέλφων που βρίσκονται στη Βαγδάτη, στο Ερμπίλ. Δεν αποκλείεται όμως κάποια χρονική στιγμή να μπορέσουν οι πολιτικές αρχές μας, να κρίνουν οι πολιτικές μας αρχές ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιος παρόν σε πλήρη χρόνο στο Ερμπίλ, γιατί είναι σημαντικοί οι συνομιλητές μας στο Ερμπίλ και όπως είπα πρέπει να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το ανθρωπιστικό του καθήκον. Έχουμε βέβαια την ΕΚΟ παρούσα εκεί, την ανθρωπιστική δηλαδή πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με παρόντες εκπροσώπους του Ερμπίλ τακτικά, ε, σε μόνιμη βάση, αλλά όπως είπαμε πρέπει να έχουμε και την πολιτική, την διπλωματική συνεργασία με τις αρχές των ε, Κούρδων εκεί. Τώρα για την ε, Λιβύη, μας συνθλίβει η εισαγωγή του θέματος της Λιβύης, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συγκρίνουμε με αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και το Ιράκ. Ε, προς το παρόν είναι ακόμα η κατάσταση αρκετά διαφορετική. Με όσα προβλήματα και να έχει η Λιβύη δεν συγκρίνεται με Ιράκ και Συρία. Είναι λίγες και μικρές, μικροί θύλακες που βλέπουμε από τρομοκράτες στη Λιβύη, αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ε, επιδεινωθεί κατάσταση. Για του χριστιανού ρωτήσατε εσεί εν γέννη μα απασχολεί το θέμα των μειονοτήτων, είτε πρόκειται για χριστιανού είτε για ζηδίτε, χωρί ταυτόχρονα όμω και να θέλουμε να δοθεί εντύπωση στου ε, Σουνίτε ότι όταν ε, βλέπουμε να την χάνουν μεταχείριση 10 χριστιανοί αντιδρούμε με αγανάκτηση ενώ όταν χίλιοι Σουνίτες πέφτουν θύματα κακοποίησης τότε γυρνάμε από την άλλη το βλέμμα. Δεν εννοώ ότι θα έλεγατε εσείς να υπονοήσετε κάτι τέτοιο. Απλώς έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη περιοχή με τραγική, ε, τραγικό πεπρωμένο ιδιαίτερα για αυτές τις ε, δυστυχείς μειονότητες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε σχέση με τις μειονότητες αυτές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις βοηθήσουμε. Επικοινωνούμε παραδείγματι με τις αρχές του Ερμπίλ στο Κουρδιστάν για να συζητήσουμε και θέματα των Γκεσιντή και των χριστιανών. Ιδιαίτερα στην περιοχή του όρου Σιντζάρ, εκεί που γίνανε μεγάλες σφαγές από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Για τον κύριο Οστρεβίτσιους που ρώτησε αν επηρεάζουν όλα αυτά το διάλογο για την ασφάλεια με το Ισραήλ. Κοιτάξτε, όταν γίνεται ο διάλογος για την πολιτική και την ασφάλεια με το Ισραήλ, προφανώς και συζητείται η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, γίνεται αλληλεγγύη απόψεων σε σχέση με τα τεκτενόμενα, με τα συμβάντα σε όλες τις χώρες. Προφανώς και βρίσκονται σε υψηλό σημείο στο θεματολόγιο των συνομιλιών μας με τους ε, ε, Ισραηλινούς εταίρους τα θέματα αυτά σε ποιο βαθμό ή με ποιο τρόπο συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρε του Περσικού. Κοιτάξτε, έχουμε συνεργασία στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία με τι χώρε του Περσικού. Έχουμε συνεργασία όσον αφορά τη συζήτηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών κινημάτων και εξτρεμιστικών, σουνητικών εξτρεμιστικών κινημάτων και εν γέννη ακούμε ή τις απόψεις τους, παρακολουθούμε τις θέσεις τους όσον αφορά το πρόβλημα της ε, ρίζοσπαστικοποίησης που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς. Δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω. Ανθρωπιστική βοήθεια, κυρία Σέμπαλος. Ε, η απάντησή μου θα είναι ότι δεν είναι ευχερής η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους πολίτες. Καταρχάς για τη Συρία γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα που ονομάζεται cross-line και cross-border. Εμείς προσπαθούμε με βάση τα ε, ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας να διοχετεύσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις προσπάθειες του Στάφαν Μιστούρα. Αυτό προσπαθεί να διαπραγματευτεί μεταξύ άλλων με τις αρχές της Δαμασκού. Υπάρχουν όμως εμπόδια και από τις δύο πλευρές και κυρίως από το καθεστώς του, ε, του Ασάτ της Δαμασκού που θέλει να εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια μεταξύ άλλων η ιδεολογική διάσταση τώρα και οι νέοι μαχητές από τις χώρες μας που πάνε στα κινήματα αυτά, τα βαρβαρι... κάνουν αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Νομίζω ότι υπάρχει δουλειά ιδεολογική που θα πρέπει να αναπτύξουμε αν θέλουμε να σταματήσουν να πηγαίνουν αυτοί οι νέοι. Πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλάμ και ότι οι στόχοι τους δεν μπορούν να βρουν απολογία σε κανένα επίπεδο ε, αυτός είναι ο αγώνας μας, αυτός είναι ο αγώνας που ξεκινάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ο Ζιλντε Κέρκοφ εδώ και μήνες κάνει πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά στον τομέα αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, αλλά και με τα κράτη εταίρους από την ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας και του ελέγχου στα σύνορα ε, και την ε, προσπάθεια να εντοπίζονται πιο πρόωρα. Οι πηγές εκείνες, ε, οι λόγοι αυτοί που προσελκύουν τους νέους να πάνε στα κράτη αυτά, να αγωνιστούν για κάποια ιδεώδη, μέσα βέβαια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έτσι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη δύναμη έλξης που μπορεί να ασκούν αυτά τα εξτρεμιστικά κινήματα σε νέους ε, που έχουν κάπως χάσει τον μπούσουλα. Για το Ιράκ, δεν έχω να διαβάσω κανένα, καμία κρυστάλλινη μπάλα. Ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του Ιράκ, τι πρέπει να γίνει ώστε να μην διαλυθεί και να μην επιδεινωθεί το, γενικό, το γενικευμένο χάος. Για τον κύριο Καν και τις Ηνωμένε Πολιτείες που με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια υποτίθεται ότι εκπαίδευσαν Ιρακινό στρατό και την ερώτηση αν θα μπορούσαν αυτή τη φορά να έχουν περισσότερη επιτυχία. Ε, κοιτάξτε τώρα με το Ιράκ. Αυτό που συνέβαινε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ο Πρωθυπουργό Μαλική είχε μετατρέψει τον στρατό, τον εθνικό στρατό, σε σιητική πολιτοφυλακή. Ε, τι έγινε λοιπόν, οι Σουνίτε αποχώρησαν από το στράτευμα και αυτό σε μεγάλο βαθμό εξηγεί τα όσα συνέβησαν γύρω από την περιοχή της Μοσούλης όταν το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος μπήκε και κατέλαβε μεγάλο μέρος της ε, Μοσούλης και αυτό σημαίνει βεβαίως, εξηγεί μάλλον καλύτερα και γιατί απέτυχε ο Ιρακινός στρατός στη Φαλούσα και στη Ράνβα. Ε, η δουλειά λοιπόν των Αμερικανών δεν ήταν περίτη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν άχρηστη. Αλλά ακυρώθηκε, ματαιώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική προτίμηση συγκεκριμένου δόγματος του Πρωθυπουργού Αλμαλίκη μέχρι τώρα. Άρα τώρα η όποια δουλειά κάνουν οι Αμερικανοί και οι λοιποί θα πρέπει να παρακολουθηθεί, να συνοδευτεί από μια πιο ανοιχτή προς όλους τους πολίτες του κράτους της νέας κυβέρνησης του Ιράκου, που εμείς δεν μπορούμε να εμπλακούμε. Τουρκία και τι κάνουμε εσείς με την Τουρκία. Προφανώς πρέπει να εντείνουμε το διάλογο με τους Τούρκους, πρέπει να προσπαθήσουμε να τους εξηγήσουμε ότι έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα. Ένα πρώτο κοινό συμφέρον ασφαλώς είναι η αποδιάρθρωση το δυνατό του λεγόμενου τελικού κράτους που αποτελεί σε πρώτο, σε πρώτο βαθμό ε, πρόβλημα και απειλή για την ίδια την Τουρκία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις αρχές της Τουρκίας για να διευκολύνουμε τη μετάβαση, μία μετάβαση στη Συρία που θα οδηγήσει σταδιακά προ μία κυβέρνηση που θα ανταποκρίνεται στις νόμιμες, στις θεμητές προσδοκίες του, ε, του Συριακού λαού και που θα μπορέσει να αποτελέσει έτσι ένα γείτονα ειρηνικό για την ε, Τουρκία. Ε, για δε το Ιράκ νομίζω ότι συμφωνούμε ότι θέλουμε ένα ενιαίο Ιράκ, ένα Ιράκ δημοκρατικό, ένα Ιράκ με κράτος δικαίου. Αυτά νομίζω ήταν εν ολίγης οι απαντήσεις ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα, πολύ ολοκληρωμένα. Θα ήταν ίσως χρήσιμο για μας ε, να μας πείτε δύο λόγια για την διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας ε, εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ. Γιατί εμείς ε, έχουμε κάνει τα απαραίτητα, αλλά πρέπει να μα πείτε τι συμβαίνει και σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο αριθμό κρατών μελών, δεν, μπορώ, δεν ξέρω όμω πόσο ακριβώ, που δεν έχω ακόμα κυρώσει αυτή τη συμφωνία. Μεταξύ 5 και 10 είναι αυτά τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, κυρώσει την ε, συμφωνία συνεργασία. Το υπερθυμίζουμε συστηματικά. Και θα είναι κρίμα να μην μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πλήρω αυτή τη συμφωνία εξαιτία τη ε, μη κύρωσης από κάποιες ε, χώρες. Ενώ το κοινοβούλιο ε, του Ιράκ το έχει ήδη κυρώσει εδώ και αρκετό καιρό. Ωραία. Δεν έρθει ο κύριος Βημών για την συζήτηση στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να επισημάνω τη δημιουργία μια συγκεκριμένη αφήγηση από πλευρά ε, υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά ε, τον πόλεμο των media για τον ISIS. Το μηντιακό πόλεμο μάλλον που κάνει και το ISIS. Ήταν ε, ιδιαίτερα δραστήριοι και είχαν και συγκεκριμένες επιτυχίε σε ό,τι αφορά του αλλαδοπούς μαχητέ και νομίζω ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη η προσέγγιση μα και ισχυρή. για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, τάσει που παρακολουθήσαμε τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαγκαρίνη για την ε, σύνοψή σας. Είστε επανειδήν. Ευχαριστώ. Uh, dear colleagues, we will just... Συνάδελφοι, λίγη υπομονή ακόμα, 5-6 λεπτά και θα έρθει ο κύριος Βημόν για να κάνουμε την ενημέρωση για τις Σημερινέ διαβουλευσει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν. Ευχαριστώ. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω τον κύριο Πιάγ με βοηθός Γενικό Γραμματεία της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, αργοπόρησε λίγο, αλλά και το Συμβούλιο άργησε τις εργασίες του. Μετά την ε, εκ των προτέρων ενημέρωση της κυρίας Μογκερίνη που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα έχουμε την ε, κανονική ενημέρωση ε, για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά. Όλοι ξέρετε την μέσα διάταξη. Αύριο η συζήτηση θα εστιαστεί στα ζητήματα άμυνα. Επομένω, δεν θα εξετάσουμε τώρα αυτό το σημείο, αλλά θα συζητηθεί και στην αφέτια στις ένα εν χρόνο. Είναι σημαντικό για μας να ακούσουμε τις βασικές πτυχές της συζήτησης ε, για την Ουκρανία. Γιατί και εμείς το συζητήσαμε σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, κύριο Κλίμκιν, και θα θέλαμε να μας πείτε και τα τελευταία νέα σχετικά με την ενεργητική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τα συμπεράσματα, ε, την τελική απόφαση για τον έμπολα. Κάτι πολύ σημαντικό που θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια την μόνη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στρασβούργο. Υπήρξε συζήτηση και για την κατάσταση στη Βοσνία και Ερσεγοβίνη μετά τις εκλογές που έγιναν στις 12 Οκτωβρίου. Και τώρα σχηματίζεται κοινοβούλιο, υπάρχει νέος πρόεδρος. κατόπιν ε, πρωτοβουλία του Γερμανού και Βρετανού Υπουργού. Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε θίξει, κάτι που συνδέεται με την Ανατολική Ευρώπη. Ε, παρακολουθούμε στενά την ε, ε, συζήτηση ε, στην Σερβία. Ο Βόσλαβ Σέζελ, εγκληματίας πολέμου, έχει ε, απελευθερωθεί και προσπαθεί να θέσει και πάλι στο δημόσιο διάλογο όλη αυτή τη ρητορική του πολέμου με περαιτέρω φιλοδοξίες για τη Μεγάλη Σερβία. Και αυτό χρήζει καταδίκης και από το Συμβούλιο αλλά και από το Ευρωκοινοβούλιο. Τέτοιου είδους συμπεριφορές ε, δεν μπορούμε να τις ε, δεχθούμε. Και πάλι πρόκειται βεβαίως για προσωρινή απελευθέρωση, αλλά και πάλι είναι εντελώς δυσανάλογο με τα όσα έχουμε δει ε, ως τώρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Βημό και μετά να περάσουμε σε συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πάλι ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά όπως αναφέρθηκε... Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, άργησε να ολοκληρωθεί. Πριν από 10-15 λεπτά τελείωσε και είπατε εκπρόσωπος ακόμα κάνει αυτή τη στιγμή την συνέντευξη τύπου. Να διατρέξω εν συντομία τα διάφορα σημεία ε, της μέσας διάταξης. Όπως ξέρετε, το πιο σημαντικό αφορούσε την Ουκρανία. Αποφασίστηκε να αποτελέσει το κύριο σημείο της πολιτικής συζήτησης ε, αυτή τη φορά. Όπως ξέρετε, θέλουμε να δοκιμάσουμε ένα νέο τρόπο διοργάνωσης αυτών των ε, συνεδριάσεων, του Συμβουλίου δηλαδή Εξωτερικών Υποθέσεων, με, δίνοντας κάθε φορά ιδιαίτερη έμφαση σε ένα από τα σημεία που απασχολούν τους Υπουργούς Εξωτερικών. Αυτό το μήνα είχαμε την Ουκρανία, την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρουμε ακόμα, ίσως Συρία ή Ιράκ, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Επομένω, η πρωινή συνεδρίαση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την Ουκρανία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, το δίχως άλλο, και στο τέλος ο είπατε εκπρόσωπος προσπάθησε να συνοψίσει τη συζήτηση ε, μέσω ορισμένων πολιτικών συμπερασμάτων. Και πλέον πρόκειται για συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα δείτε ότι θα ε, δημοσιευθούν μέσα στα επόμενα λεπτά. Τα δικά της πολιτικά συμπεράσματα είναι ότι όλοι συμφωνούμε πως είμαστε αντιμέτωποι με μία μείζον ευρωπαϊκή κρίση στην Ουκρανία και επομένως και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι διπλωματικά δραστήρια σε αυτή την κρίση, ίσως και περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Να είμαστε λοιπόν ενεργοί και δραστήριοι ως προς την Ουκρανία και ως προς τη Ρωσία. Υπογράμμισε επίσης ότι είναι σημαντικό να ε, αναφερόμαστε συνεχώς στο πρωτόκολλο Μίνσκ, όπως, καθώς είναι το μοναδικό συμπεφωνημένο κείμενο σήμερα, και ίσως πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση, μια νέα δυναμική στις προσπάθειες ε, που καταβάλλονται αυτή τη στιγμή, ε, κυρίως στις προσπάθειες του ΟΑΣΕ, με την τριμερή ομάδα επαφών ε, που ε, συνεδριάζει στο Μίνσκ ε, ανατάκτα χρονικά διαστήματα και θα δώσουμε την πλήρη στήριξή μας. Ανέφερε επίσης κάτι που υπήρχε και στο αρχικό κείμενο που είχαμε επιτάπητος, δηλαδή οι προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κατευθύνονται αφενός προς την επαναφορά της ειρήνης ε, στην Ανατολική Ουκρανία με ό,τι συνδέεται με την εφαρμογή του εγγράφου του Μίνσκ κατά πυρός, ε, διαχωριστική γραμμή ε, μεταξύ των δύο πλευρών, αποστολή παρακολούθησης του ΟΑΣΕ, εφαρμογή ελέγχων μεταξύ ε, Ρωσίας και Ουκρανίας, ανθρωπιστική αρρωγή και πολλοί ανέφεραν ότι καθώς ε, πλησιάζει και ο χειμώνας, μπορεί να αυξηθούν οι ροές προσφύγων στη Δυτική Ουκρανία αλλά και ενδεχομένω και σε άλλες ε, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέραν της Ουκρανίας δηλαδή. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση και ως προς αυτό το ζήτημα. Και να δούμε πώς μπορούμε να πείσουμε και τη Ρωσία να τηρήσει, να σεβαστεί το πρωτόκολλο Μίντσκ. Ε, με την ε, απόσυρση ε, είτε στρατιωτικού εξοπλισμού είτε ακόμα και στρατιωτικών δυνάμεων και δεύτερον πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε όλες ε, τις πλευρές ε, του πρωτοκόλου του Μίνσκ. Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε τη στήριξη προς την Ουκρανία στην πορεία της ε, προς τη μεταρρύθμιση. Και εδώ έχουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που καλύπτονται από την Συμφωνία Σύνδεσης, κάτι που αφορά κυρίως τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, πώς θα εφαρμόσουμε το κράτος δικαίου στην Ουκρανία. Και, θα και πώς θα δώσουμε ε, τις δυνατότητες, απαραίτητες δυνατότητες στις Ουκρανικές αρχές για να υιοθετήσει και να εφαρμόσει την νομοθεσία στον δικαστικό τομέα, στο μέτρο ενέργεια και το καθεξής. Πολλά ενέφεραν ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα της συνταγματικής διαδικασίας που ανέκυψαν πριν από το καλοκαίρι και φαίνεται ότι έχουν χάσει κάπως τη δυναμική τους. Με τον όρο συνταγματική διαδικασία εννοούμε οτιδήποτε συνδέεται με την αποκέντρωση με ε, το καθεστώς ε, των μειονοτήτων, των ρωσόφωνων μειονοτήτων, εκλογική μεταρρύθμιση και το καθεξής. Θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Βέβαια, για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μια νέα ουκρανική κυβέρνηση και από όλα τα κράτη-μέλη υπάρχει η αίσθηση ότι θα πρέπει να ε, παρακινήσουμε τις ουκρανικές αρχές να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις συζητήσεις για, το, για τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού και έτσι να σχηματιστεί όσο γίνεται πιο γρήγορα νέα κυβέρνηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ο χρόνος εδώ. Και το τρίτο μέρος των συζητήσεων αφορούσε το πώς ενώ θα είμαστε και ανοιχτοί ε, προς ένα διάλογο με τη Ρωσία, παρά τα όσα συμβαίνουν επί τόπου, υπάρχει ανάγκη να είμαστε αμετακίνητη και να υπενθυμίζουμε στη Ρωσία ότι ε, αν δεν υπάρξει βελτίωση θα πρέπει να περάσουμε σε νέες κυρώσεις. Σε αυτή τη φάση οι Υπουργοί αποφάσισαν σήμερα να ζητήσουν από το Συμβούλιο, κυρίως ε, την Κορεπέρ, ε, σε επόμενες εβδομάδες, πριν τα τέλη του μήνα δηλαδή, να έχουν έναν επιπρόσθετο κατάλογο για τους ε, Ρώσους αποσχιστές. Ε, μετά τις ε, εκλογές στην Ανατολική Ουκρανία, τις οποίες εμείς κηρύξαμε παράνομες και μη αποδεκτές, αποφασίσαμε σήμερα να υπάρχουν και νέα ονόματα στον κατάλογο των ατόμων που υπόκειται σε κυρώσεις, είτε με το πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων, είτε με ε, απαγόρευση εισόδου και θεώρησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα δράσουμε, θα ενεργήσουμε όπου δει. Και πάλι υπάρχει το ενδεχόμενο να καταφύγουμε σε οικονομικές κυρώσεις, αλλά προς το παρόν δεν κάνουμε κάτι. Και υπήρξε και ζήτημα για την Κρυμαία. Παραβιβαιώσαμε την άρνησή μας, την απόρριψη οποιασδήποτε προσάρτησης της ε, Κρυμαίας. Ξέρετε ότι και πρόσφατα είχαμε αποφασίσει εμπορικές και επενδυτικές απαγορεύσεις και κυρώσεις σε ό,τι αφορά συγκεκριμένους ε, κλάδους, ενέργεια, μεταφορές και το καθεξής. Θα δούμε τι θα χρειαστεί να γίνει στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα το εξετάσουν. Αυτά για την Ουκρανία. Μετά είχαμε το γεύμα, όπου συζητήσαμε την ενευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Όπως είπατε, Πρόεδρε, έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου, υιοθετήθηκαν μετά το γεύμα. Στο γεύμα, κυρίω ε, είπατε εκπρόσωπο και κάποιοι υπουργοί μίλησαν, είχαν ε, επισκεφθεί την περιοχή. Μοιράστηκαν λοιπόν τις εντυπώσεις τους από αυτή την επίσκεψη. Δύο-τρία βασικά σημεία. Αρχικά, η εγχώρια πολιτική σκηνή και στις δύο πλευρές ήρθαν στο προσκήνιο, δηλαδή γενικές εκλογές που σιγά σιγά πλησιάζουν στο Ισραήλ, ε, που ε, δυσκολεύουν έτσι την Ισραηλική κυβέρνηση να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. Και έτσι ευθυγραμμίζεται όλο ένα και περισσότερο από τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία του συνασπισμού και από την άλλη σημαντική δυσκολία αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Παλαιστινιακή πλευρά. Δυσκολεύεται λοιπόν να καλύψει τα βασικά ζητήματα που αφορούν την Παλαιστινιακή Αρχή και τη Χαμάς. Παρά το γεγονό ότι επισκεφθήκαμε την, ε, τη Γάζα πριν από ε, μερικές εβδομάδες, διατηρείται αυτός ο διχασμός και έτσι τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορούμε δυστυχώς ε, να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. οι συζητήσεις και σε, στην περιοχή αλλά και στην Νέα Υόρκη αφορούν την προοπτική ενός νέου ψηφίσματος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή και προωθείται από την Πολυστινιακή Αρχή. Ένα τέτοιο ψήφισμα θα έθετε μια προθεσμία για την αναγνώριση της Παλαιστινιακής Αρχής στις, ε, στην κατεχόμενη επικράτεια της Γάζας ως ε, οριστική απόφαση. Το βασικό ζήτημα για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος είναι αν θα συγκεντρώσει τις απαραίτητες εννέα ψήφους και αν τις συγκεντρώσει είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξει βέτο από τουλάχιστον ένα από τα πέντε μεγάλα μόνιμα μέλη. Και έτσι πώς ε, θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε και πώς θα πείσουμε την Παλαισθενική Αρχή να τροποποιήσει ε, το ψήφισμα ε, για να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και το τρίτο θέμα βεβαίως αφορά ε, την διάχυση των γεννήσεων μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, τη διάδοση μάλλον αυτή τη τάση ε, αναγνώριση τη Παλαιστινική Αρχή, όπω έχουμε δει και στην Σουηδία, αλλά και ήταν απόφαση τη κυβέρνηση, αλλά και πιο πρόσφατα και στο Λονδίνο. Και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και στην Ισπανία, στη Γαλλία και σε άλλα κράτη-μέλη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, παρενέβησαν για να επισημάνουν ότι ε, προδιαγράφεται μια τέτοια πορεία και στη χώρα τους. Κάποιοι από τους υπουργούς τα ανέφεραν τουλάχιστον. Μετά το γεύμα έγινε μια σύντομη συζήτηση για τον έμπολα. Ο Επίτροπος κ. Τελιανίδης ε, που επέστρεψε από την ε, Αφρική και την περιοδία που έκανε εκεί και επεσήμανε ότι η κατάσταση εκεί είναι ακόμα ιδιαίτερα ε, ρευστή. Ιδίως στην Ιγυρία όπου μάλλον εκτός από την Νιγηρία όπου ε, ο αριθμός των ασθενών σταθεροποιείται, στην Σιέρα Λεόνη και στην Κινέα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολλοί φοβούνται ότι θα ε, χειροτερεύσουν τα πράγματα μέσα στις επόμενες ημέρες, γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο ιατρικό προσωπικό, περισσότερες ε, δυνατότητες εκένωσης, εάν αυτό χρειαστεί, και σίγουρα οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν. Η τέταρτη μνήμα έγινε στην πρωτοβουλία ε, Γερμανίας και Γαλλίας να συστήσουν ε, τη δύναμη των λεγόμενων ε, λευκόκρανων. Όλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για μια θετική πρωτοβουλία, αλλά αναφέρθηκε ότι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος να υπονομευθούν οι φυστάμενες προσπάθειες από την ανάγκη να συζητήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν να το εξετάσουμε, να εξετάσουμε αυτή την νέα πρωτοβουλία ε, σε ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα ε, από τα όσα εξετάζονται για τον έμπολα. Για τη Βοσνία, πρόεδρε, ορισμένοι υπουργοί αναφέρθηκαν στις δηλώσεις ε, του πολιτικού ηγέτη αυτής της χώρας και πολλοί είπαν ότι θα πρέπει να ε, κάπως να απαντήσουμε. Η συζήτηση κυρίως αφορούσε ε, την τελευταία πρωτοβουλία Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή ένας νέος τρόπος προσέγγισης του ζητήματος της Βοσνίας και συνέχιση της εφαρμογής των προϋποθέσεων που ζητούμε από τις ε, βοσνιακές αρχές. Αντί λοιπόν να έχουμε μια προϋπόθεση, απαραίτητη ε, προϋπόθεση χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πρέπει να δώσουμε μια νέα δυναμική στην όλη διαδικασία και γι' αυτό με την επίδειξη κάποιας εμπιστοσύνης να πιέσουμε, να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τους πολιτικούς ηγέτες της ε, χώρες αυτής για να κινηθούν προς τις ε, μεταρρυθμίσεις που επιθυμούμε. και στην πορεία να αξιοποιήσουμε τη μόχλευση ολόκληρης διαδικασίας ε, διεύρυνσης για να διαμορφώσουμε έναν κύκλο, ευρύτερο κύκλο, που θα βοηθήσει και αυτή τη χώρα να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη δουλειά για να δούμε πώ ακριβώς θα γίνει αυτή ε, η αλληλουχία κινήσεων. Οι πρέσβεις του PCSC θα μεταβούν στη Βοσνία μέσα τι επόμενε ημέρες και μετά θα εξετάσουμε με ποιον τρόπο ακριβώ θα εργαστούμε. Τέλο ε, Βοσνία και κλείνω εδώ, όλοι συμφωνούν ότι η κατάσταση γίνεται λένε και πιο δύσκολη. Όπως ξέρετε υπήρξε ακόμα και το ενδεχόμενο ε, συνδιάσκεψη στη Μαδρίτη μέσα σε δύο ημέρες που από, πάνω από 22 χώρες θα μπορούσαν να είχαν εξετάσει την κατάσταση. Τελικά όμως αποφασίστηκε να αναβληθεί η διάσκεψη γιατί ακόμα είναι ρευστή η κατάσταση. Όλοι όμως συμφώνησαν να μείνουμε στην προσέγγιση ότι στηρίζουμε ε, το Μπερναντίνο Ντελεόν, ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ, και ουσιαστικά προσπαθούμε να προαγάγουμε τον δημόσιο διάλογο, τον εθνικό διάλογο σε αυτές τις χώρες ε, βάσει και των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λιβύης που διακήρυξε άκυρες ε, τις πρόσφατες ε, κοινοβουλευτικές βουλευτικές μάλλον εκλογές και γι' αυτό θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο εθνικό διάλογο. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή γιατί κάποια κόμματα δεν έχουν καθόλου επαφές μεταξύ τους και προσπαθούν να αξιοποιήσουν στρατιωτικά μέσα για να επιβάλλουν ε, την άποψή τους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, τρόπο να συγγύσουν αυτά τα όπλα και να ξανακαθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων όλες αυτές οι πλευρές. Αποφασίστηκε τελικά οι Υπουργοί να επανέλθουν σε αυτό το ζήτημα το τών. δυνατόν, γιατί ακόμα μένουν πολλά να υποθούν και εν μεταξύ θα προσπαθήσουμε να θέσουμε ε, σαφείς και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις επιτάπητος για να δούμε τι μπορεί να κάνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί να συμβάλλει στις προσπάθειες του ΟΗΕ. Θα μείνω εδώ να προσθέσω μόνο ότι ε, σήμερα στο πρόγευμα υπήρξαν συζητήσεις για τη μέθοδο λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών Υποθέσεων Όπω ανέφερα και προηγουμένω, θα πρέπει να επικεντρώνεται κάθε ε, συνεδρίαση σε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα, να έχουμε μικρότερη μέσα διάταξη, με καλύτερη προετοιμασία, με συγκεκριμένα έγγραφα και προσχέδια συμπερασμάτων, τα οποία θα ε, διαβιβάζονται στι αντιπροσωπείε εκ των προτέρων, για να υπάρχει δυνατότητα προετοιμασία από εκείνου. Ίσως μπορούμε να οργανώνουμε με καλύτερο τρόπο τη συζήτηση για να είναι πιο ζωντανή ε, η συζήτηση με καλύτερο πολιτικό προσανατολισμό, αλλά και με καλύτερα αποτελέσματα. Με γνώμονα δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα. Όλοι συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, όλοι ε, ήταν μάλλον επιφυλεκτικοί για το κατά πόσο θα πετύχουν αυτές μας οι προσπάθειες, γιατί το κύριο σημείο τελικά είναι ο χρόνος. Δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους, μία φορά το μήνα μερικές ώρες, επομένως πέραν οποιασδήποτε προσθήκης ε, ε, στο Συμβούλιο Ευθυνικών Υποθέσεων μπορεί να έχουμε και άλλες συνεδριάσεις ε, άτυπες. Θα επανέλθουν σε αυτό τον επόμενο μήνα σε μια άλλη άτυπη συνεδρίαση για να δούμε αν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την προσέγγιση για τον τρόπο λειτουργίας. Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ. Ανοίγουμε εδώ τη συζήτηση. Ο Αλόης Πέτερλε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας των συμπεράσματων στο Συμβούλιο σήμερα. Με χαρά άκουσα όχι μόνο για τη μέθοδο εργασίας, αλλά πρώτα απ' όλα για δύο κέντρα βάρους σε σημαντικά θέματα που προάγονται αυτή τη στιγμή. Το ένα σε σχέση με την Ουκρανία, το άλλο σε σχέση με την Βοσνία. Θα έλεγα ότι το κέντρο βάρους στις μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικό θα ευχόμουν ιδιαίτερη προσοχή να δίναμε, να δινόταν στην χρηστή διαχείριση, διακυβέρνηση, όχι μόνο για το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και πολλών άλλων χωρών επίσης, που είναι εταίροι μας και που θα έλεγα διαρκής μόνιμη προσοχής, μόνιμης προσοχής πρέπει να την χάνουν και σύνδρομης και βοήθειας. Με ικανοποίησε επίσης αυτό το οποίο αναφέρθηκε ότι συζητήθηκε σήμερα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη σχετικά. Και πιστεύω ότι πραγματικά ήρθε η χρονική στιγμή να δράσουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μετά από τόσα πολλά χρόνια που δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος ή μάλιστα κιόλα επιδεινώθηκε η κατάσταση εκεί και πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω, περισσότερο εκεί και μου άρεσε αυτό το οποίο περιγράψατε. <clears throat> Σε σχέση με όσο λιγότερο εμπλεκόμαστε ή εμπλέκεστε εσείς τόσο περισσότερο θα εμπλέκονται άλλοι και δεν θα ευθυγραμμίζονται καθόλου και με τα συμφέροντά μας σε αυτή τους την προσπάθεια. Αναμένω λοιπόν κάτι να υπάρξει όπως η φιλοδοξία που καταδείχθηκε στην περίπτωση του διαλόγου μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Και εδώ πάλι πρέπει να καταδειχθεί κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε περισσότερα στοιχεία βέβαια, αλλά έχουμε θετική πείρα με αυτό το διάλογο που προανέφερα και θα έλπιζα η δράση, η κίνηση να στοχεύει προς την κατεύθυνση που περιγράψατε σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Uh, θα σε ευχαριστώ. Και σε σχέση με την ε, παρέμβαση αυτή θέλω να ευχαριστήσω. Πολύ θετικές ε, οι συζητήσεις με την κυρία Μογκερίνη και για την ε, επόμενη περίοδο τα όσα προβλήματα. Τρεις παρατηρήσεις για την Ουκρανία. Μια σύντομη ε, σύγκριση σε όσα είχαν συμφωνηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα συμπεράσματα. Και είναι δραματική κατάσταση σε σχέση με τα όσα περιγράφονται. Πρέπει ταχύτατα να υπάρξει δράση ε, είναι μια καμπή αυτή, μια νέα προσοχή, μια νέα κατάσταση πραγμάτων αναδύεται εκεί σε σχέση με τα όσα υπήρχαν κατά το παρελθόν. Και η περιγραφή των όσων συνέβησαν είναι νομίζω και αυτό ε, σημαντικό στοιχείο. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερα δραματικό, ιδιαίτερα σε σχέση με την προσπάθεια να δοθεί μια νέα όθηση σε σχέση με συνταγματικά θέματα και δικαιώματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, είμαι λοιπόν ε, ευγνώμων ε, για, την, το σχόλιο σας επ' αυτού και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν το, σήμερα το απόγευμα για την προπαρασκευή μέτρων κατά των αποσχιστικών τάσεων και σε σχέση και με τις παράνομες αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις ε, όσον αφορά την, ε, τα εδάφη, την επικράτεια της Ουκρανίας. Διαρωτώ με, πώς αυτά τα δύο ε, συνάδουν και συνδέονται όσον αφορά και τα θέματα κυρώσεων για το θέμα της Παλαιστίνης. Μπορείτε να αποσαφηνίσετε παρακαλώ σε σχέση με τους Υπουργούς Εξωτερικών για το θέμα της αναγνώρισης, ε, για παράδειγμα, κάποιων κρατών που έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη από πλευράς κοινοβουλίων, που βρίσκονται οι κυβερνήσεις σε σχέση με την ε, προώθηση αυτής της ε, τάσης αναγνώρισης των Παλαιστινίων, του Παλαιστινιακού κράτους και δεδομένη τη επίσκεψη τη κυρία Μογκερίνη σε αυτή την περιοχή, υπήρξαν κάποια σχόλια που έγιναν σε σχέση με του Παλαιστίνιου. Ποιο ήταν ο τόνο και η απάντηση, ο τόνος στον οποίο εκφράστηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών σε σχέση με αυτό το θέμα και σε σχέση με το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνη, μια τελευταία παρατήρηση. Θα έλεγα ότι νομίζω ότι αυτό το οποίο άκουσα είναι ότι θα επανέλθει λέει το Συμβούλιο επ' αυτού. Υπάρχει και η Αγγλογερμανική πρωτοβουλία σε σχέση με την ε, ε, κατάσταση εκεί. Υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε, τροποποιήθηκε η Αγγλογερμανική πρωτοβουλία. Υπήρξε περαιτέρω συζήτηση αυτού του θέματος. Ποιο είναι το καθεστώς αυτής της ε, Αγγλογερμανικής πρωτοβουλίας υπό το φως των συναντήσεων του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαουίτς. Τώρα ο κύριος Ντεμέσμακερ παρακαλώ. Ε, ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Βημό για την ενημέρωση. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω στο ζήτημα της Ουκρανίας. Έχω μερικά ερωτήματα από αυτού. Είπατε ότι κατά το Συμβούλιο θα πρέπει κάτι να γίνει για τους πρόσφυγες. Νομίζω είναι 400.000 IDPs, δηλαδή ε, εσωτερικά εκτοπιστέντες. Αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο που εγώ άκουσα για την Ουκρανία. Το καλοκαίρι ήμουνα στον ιέτρο Πετρόφσκ και Εκείνη τη στιγμή κιόλα ήταν χιλιάδε τα άτομα που έφταναν ε, στην περιοχή και ήταν σαφέ ότι εκατοντάδε χιλιάδε θα χρειαζόντουσαν βοήθεια. Οι τοπικέ αρχέ είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πέρασε και το καλοκαίρι, ξεκίνησε ο χειμώνα και πολλοί από αυτούς ε, έχουν ε, δύσκολους καιρούς μπροστά τους. Αν δεν λάβουν την απαραίτητη βοήθεια, πράγματι θα εμφανιστούν στις πρωτεύουσές μας. Θα στραφούν προς εμάς. Και τι θα γίνει τότε. Επομένω, το ερώτημά μου είναι, όταν λέει το Κοινοβούλιο κάτι πρέπει να γίνει, τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα, πόσο γρήγορα θα αντιδράσουμε ε, και πόσο συγκεκριμένα. Για την Κρυμαία, η ιδέα της ε, προσάρτησης απορρίπτεται. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί και το Συμβούλιο κατανοεί ότι όταν υιοθετούνται οικονομικά ε, μέσα, πρέπει να αναλογίζεται ότι και κατάσταση, η οικονομική κατάσταση των ε, ε, κατοίκων είναι εξαιρετικά αρνητική. Έχουμε πολύ ανησυχητικά φαινόμενα, εξαφανίσεις, δολοφονίες. είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί και θα κάνετε κάτι. Και τέλος, δεν θα υπάρξουν οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία, ούτε το ανέμενε κάποιος αυτό νομίζω. Το Συμβούλιο εννοεί ότι οι υφιστάμενες ε, οικονομικές κυρώσεις είναι επαρκείς, είναι κατάλληλες, είναι επιτυχείς και θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη ρωσική πλευρά, πλευρά προς ε, μια πιο επικοδομητική προσέγγιση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you, Mark. Ευχαριστώ, Μάρκ. Τώρα ο λόγος στον Έντουαρτ Κουκάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Πρόκειται για μια ρεαλιστική προσέγγιση που την εκτιμώ μου πολύ. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε ένα ζήτημα, στην Βεσνή και ο Ζεγοβίνη. Χάρηκα που άκουσα ότι το Συμβούλιο αφιέρωσε πολύ χρόνο στην πρωτοβουλία των Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας και Ηνωμένου Βεσιλείου. Μελέτησα την επιστολή τους προσεκτικά και φαίνεται ότι πρόκειται για μια πραγματικά θαραλέα πρωτοβουλία με πολλές καινοτόμες ιδέες, με πολλές ε, νέες ε, ε, προϋποθέσεις, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είδα επίσης ότι δεν πρόκειται για μια πρωτοβουλία μεταξύ των δύο αυτών χωρών, αλλά και ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ε, απέδωσε μεγάλη ε, σημασία σε αυτό. Για την Βοσνία ε, Ερζεγοβίνη, νομίζω ότι πρέπει να εξηγηθεί διεξοδικά ότι πρόκειται για μια νέα ευκαιρία για εκείνους, για το πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά εκείνοι και θα πρέπει έτσι να αντιληφθούν την πρωτοβουλία αυτή, διότι αν αυτή η πρωτοβουλία που πραγματικά νομίζω ότι ε, χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Αν αποτύχει λοιπόν τότε ε, δεν ξέρω τι, πρόκειται, τι άλλο πρόκειται τελικά να δώσει όθηση προς, το, προς τα εμπρός ε, στη, στη χώρα. Δεν ξέρω ε, τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε για να εξηγήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα και την θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει βοήθεια και υπηρεσίες προς τη χώρα αυτή. Οπότε αυτό που είπατε ακούγεται πολύ ενθαρρυντικό, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Έντουαρτ. Ο λόγος στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Βεμόν, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ο συνάδελφος Ρίτσαρτ σας ρώτησε ήδη για την επίσκεψη της ε, είπα της εκπροσώπου στην Λωρίδα της Γάζας. Μπορείτε εσείς να μας πείτε αν υπάρχουν ε, επιπτώσεις ε, στην δήλωσή της από τα όσα είδε και από τα όσα συζήτησε εκεί είναι κάτι που περιμένετε να μετουσιωθεί και σε μια πιο επιταχυμένη διαδικασία αναγνώρισης της Παλαιστίνης. Είπατε ότι το περιμένετε, αλλά θεωρείτε ότι πραγματικά θα αποτελέσει τμήμα μιας διαδικασίας που θεωρεί η κυρία Μογκερίνη ότι θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο στις συνομιλίες της στην ε, Γάζα. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι για τη Λιβύη. Ε, αναφερθήκατε στις προκλήσεις που σχετίζονται με την απόφαση του δικαστηρίου. Υπάρχει ο κύριος Ντελεόν ως ε, ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ και φυσικά δεν με εκπλήσει καθόλου. Δεν είναι δική μας ευθύνη βέβαια. Ε, είναι και δική μας ευθύνη, όχι, όχι μόνο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών που αρνήθηκαν να δράσουν συντονισμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση ως προς την ασφάλεια που δεν επηρεάζει μόνο τον κόσμο, τους ανθρώπους στη Λιβύη, αλλά θα επηρεάσει και σε εμά σε λίγο καιρό θα έχουμε ε, θύλακες του ISIS στο έδαφος μας ε, υπάρχουν προβλήματα στην, ε, στην ε, Μάλτα, σε, σε λίγο καιρό ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα στη Μάλτα, στην Τινησία και ο Ντελεόν είναι ο μόνος που προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά, όλες αυτές τις καταστάσεις. Τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάσταση ή απλά κάθονται και σχολιάζουν την κατάσταση απ' έξω. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες και τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μιλαμόν. Ευχαριστώ. Για την κατάσταση στην Ουκρανία, δύο ερωτήσεις. Κύριε στο πλαίσιο του Συμβουλίου υπήρξε κάποιο σχόλιο, κάποια αξιολόγηση, κάποια εκτίμηση για τις επαφές ε, και τις συζητήσεις ε, στην Brisbane με αφορμή την λέσχη των 20 που είχε πάει εκεί και ο πρόεδρος Πούτιν της Ρωσίας και υπήρξαν και επαφές σε σχέση με την Ουκρανία και την κρίση στην Ουκρανία και διμερεί σε σχέση με τις επαφές τους με τον κύριο Πούτιν, ηγετών της Ευρώπης. Για την Ουκρανία η δεύτερη παρουσίαση, η δεύτερη σκέψη που θα ήθελα να παρουσιάσω σε σχέση με τα όσα είπατε. Υπάρχει από το Συμβούλιο την κυρία Μογκερίνη ε, πρόθεση να διαδραματίσει μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα όσα ε, έχουν ακολουθηθεί σε σχέση με τους Υπουργούς Εξωτερικών, ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω πέρα από την ε, κυρία Άστον σε σχέση με το τελευταίο διάστημα, υπήρχε μια βούληση νομίζω του Συμβουλίου να είναι περισσότερο παρόν το Συμβούλιο ως πολιτικά εμπλεκόμενος. Σε ποιο πλαίσιο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έγινε κάποια αναφορά στην τριμερή ομάδα επαφής Νομίζω και η ομάδα η τριμερή, δεν ξέρω ποιοι είναι και αν είναι οι αποσχιστικές δυνάμεις, οι, Ρώσοι και οι Ουκρανοί. Νομίζω αυτοί οι τρεις είναι που την συναποτελούν. Και είναι νομίζω σημαντικό αυτό το θέμα. Σαν συνέπεια αυτών η αυξημένη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως ε, εμπλεκόμενου ε, παίκτη υπό την άποψη της κυρίας Μογκερίνη, σε ποιο πλαίσιο θα διαδραματιστεί. Σε αυτή την ομάδα επαφής όπως λέγεται, όπου η Ουκρανία πιστεύω ειλικρινά ότι βρίσκεται σε μια δυσανάλογη θέση και κατάσταση, μη ισόρροπη ε, θέση σε σχέση με τη στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία και τις αποσχιστικές ε, φιλορωσικές δυνάμεις. Είναι κάπως μη ισόρροπη η κατάσταση για την Ουκρανία. Και σε σχέση με την Μέση Ανατολή για το Ισραήλ μας κάνατε λόγο για τις ε, μελλοντικές εκλογές. Όλοι ξέρουμε τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται από πλευράς του κυρίου ε, ε, Κέρικ να μπορέσει να εγγραφεί το θέμα της ειρήνευσης ε, ε, μέσα στο πλαίσιο των επόμενων εκλογών τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να κινητοποιηθεί το Ισραήλ, να αλλάξει θέσεις. Ε, θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι απόψεις της κυρίας Μογκερίνη σε σχέση με την πρόσφατη επίσκεψή της στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξουν κάποιες νέες κινήσεις το επόμενο διάστημα εκεί για κάποιες αντισταθμίσεις έχω κάποιες επιφυλάξεις. Θα ήθελα να ακούσω τι δικέ σα απόψει, τι δικέ σα εντυπωσει για τα όσα είπε η κυρία Μογκερίν μετά την επίσκεψή τη. εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Η ώρα είναι 7. Οι διερμηνείς είναι μαζί μας και μάλιστα του ευχαριστώ για όλη τη βοήθειά του για λίγα λεπτά ακόμα. Σα δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ σύντομα στα ζητήματα που τέθηκαν για την Ουκρανία. Πολλοί από εσά τονίσατε το γεγονός ότι το Συμβούλιο επέμεινε στην ανάγκη καλής διακυβέρνησης και αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο που ανέκυψε από το Συμβούλιο ε, χωρίς καμία αμφιβολία. Ακόμη και ο Επίτροπος ο κ. Χάν τόνισε ότι μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης υπάρχει μια σαφής δέσμευση για την κατάρτιση μιας ατζέντα μεταρρυθμίσεων από την Ουκρανία και ότι θα πρέπει να ε, επεξεργαστούμε έναν ε, οδικό χάρτη για τις μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα, στην ε, καταπολέμηση διαφθοράς, στην τομέα της πολιτικής προστασίας και νομίζω ότι ε, όλα τα κράτη-μέλη ε, υιοθέτησαν ε, μια προσέγγιση με βάση την οποία λέμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία. το έχουμε κάνει και οικονομικά, αλλά θα πρέπει να πάρουμε και κάποιο αντάλλαγμα. Θα πρέπει να υπάρξει πραγματική πρόοδος ως προς τις μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που προέκυψε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και νομίζω ότι αυτό κυριάρχησε σε όλη τη συζήτηση. Κύριε Χόιτ, είπατε για τις ε, νομικές δυνάμεις και τη, μήπως υπάρχει κάποια αντίφαση, ε, αν τελικά υπάρχει τίποτα καινούριο ε, στα συμπεράσματα μας. Νομίζω ότι τα συμπεράσματά μας ευθυγραμμίζονται με τα όσα έχουμε πει στο παρελθόν και ε, θα συμφωνήσετε ότι έχουμε ξανατονίσει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην ε, Ουκρανία. Για τις παράνομες δυνάμεις που υπάρχουν εκεί, επαναλαμβάνουμε αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι θα πρέπει να αποσυρθούν και επιμένουμε σε αυτό. Υπάρχει και θα το έχετε σημειώσει κι εσείς σε σχέση με όσα συνέβησαν στο Brisbane, ότι καθώς ο κύριος Προύτιν επαναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν επιθυμεί μια παγωμένη σύγκρουση στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα όμως δεν προσπαθεί να ε, λέει ότι δεν προσπαθεί να ε, θέσει σε κίνδυνο την εδαφική συνοχή της Ουκρανίας. Τα κράτη-μέλη ωστόσο εξέφρασαν την επιθυμία τους να εξεταστεί αν αυτό είναι αληθές και να ε, εξετάσουμε τις πιθανότητες να δημιουργηθεί και να οικοδομηθεί ένας νέος διάλογος με τη Ρωσία και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να, να βασιστεί στην, ε, στο, στο πρωτόκολλο του Μίνσκ. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τώρα, Ερωτήσατε για το τι εμείς θέλουμε να, τι θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό που θα είναι πιο χρήσιμο για την ε, ε, επιβολή της ε, ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτό που προέκυψε από την συνεδρίασή μας σήμερα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη υπογράμμισαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη παρουσία στις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες που καταβάλλονται αυτή τη στιγμή προκειμένου να εξευρεθεί διέξοδος από την κρίση οι τρι, τριμερείς ομάδες, η ομάδα της ε, Νορμανδίας έχετε δίκιο ε, ε στην ομάδα την τριμερή συμμετέχουν οι υποσχεστές οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί ε, έχουμε σκοπό να ε, υποστηρίξουμε την ομάδα αυτή έχουμε και άμεσες επαφές με το Κίεβο και τη Μόσχα και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στο να επανέλθουν όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί αυτή τη στιγμή η τριμερής ομάδα έχει καταφέρει να προχωρήσει και να εφαρμόσει μεγάλο μέρος των αποφάσεων που ελήφθησαν ε, στο Μίνσκ και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αναζωογονήσουμε τις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μορφή ε, στην οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, η συνάντηση της Γενέβης. Μία συνάντηση έγινε σε αυτή τη σύνθεση στις 17 Απριλίου. Είπα Ρωσία, Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν. Η Κάθριν Άστον συμμετείχε ε, σε εκείνη τη συνεδρίαση αλλά δεν έγινε ποτέ δεύτερη διότι υπόθηκε ότι οι αποσχιστές θέλουν να είναι ε, μέλος της Ουκρανικής Αντιπροσωπείας και η Ουκρανική κυβέρνηση αντέδρασε. Και θα πρέπει να δούμε εάν μπορούμε να συνεχίσουμε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η ύπατη εκπρόσωπος δεν μπορεί να έχει διμερείς επαφές. Για να γίνω στο δυνατόν πιο χρήσιμη η δική της συμβολή. Όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων, θέλω να σας δώσω ε, σαφείς συγκεκριμένους αριθμούς. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που εξέδωσε στις αρχές του καλοκαιριού ο μιλάμε για 300-400 ε, πρόσφυγες που κινούνται προς την δυτική ε, Ουκρανία και περισσότερα από 500.000 που κινούνται προς την Ρωσία, την, ε, την περιοχή του Ροστόφ και άλλες περιοχές της Ρωσίας. Και φυσικά εκφράστηκαν φόβοι ότι στη διάρκεια του χειμώνα ενδέχεται ο ρυθμός αυτός να ευξηθεί και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, ε, κάτι που μπορεί να αποτελέσει απαιτητική ανάγκη τους επόμενους μήνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους μεγαλύτερους ε, παρόχους ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε προσπαθήσει να παράσχουμε κάθε βοήθεια. Μπορούσαμε... Ε, συμμετέχει και ο Ερυθρός Σταυρός, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, συμμετέχουν και εθνικές αρχές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από τα κράτη-μέλη, έχουν ε, ε, γίνει και κάποια κονβόη. Υπάρχει λοιπόν μια δραστηριότητα, ενδεχομένως ναι, να χρειάζεται και περισσότερη. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσφυγες που έχουν ε, καταφύγει στη Δυτική Ουκρανία έχουν καταφέρει να λάβουν αρρωγή, αλλά πρέπει να, να γνωρίζουμε ότι όντως το πρόβλημα αυτό μπορεί να οξυνθεί με το πέρασμα του χρόνου. Για, το, για την Κρυμαία έχετε απόλυτο δίκιο, παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των Τατάρων, έχουμε εκφραστεί τους τελευταίους μήνες εντονότατα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και γι' αυτόν τον λόγο μεταξύ άλλων στα συμπεράσματά μας θα ε, επανεξετάσουμε τις ε, κυρώσεις κατά της Κρυμαίας για να δούμε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε ότι δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Και όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις, ναι, ε, φαίνεται ότι πράγματι είχαν κάποια αποτελέσματα και οι υπουργοί με ειλικρίνεια αποδέχθηκαν ότι δεν ήταν μόνο οι οικονομικές δυσκολίες ότι οι οικονομικές δυσκολίες της Ρωσίας δεν οφείλονται μόνο στις δικές μας ε, κυρώσεις αλλά και στη μείωση της ε, τιμής του πετρελαίου που έχει πλήξει σοβαρά την οικονομία της ε, ε, Ρωσίας και το νόμισμά της, το ρούβλι που η αξία του έχει μειωθεί σημαντικά. Προς το παρόν αποφασίσαμε ότι θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση αν χρειαστεί, αν ε, προκύψουν δραματικές εξελίξεις ε, τότε θα επανέλθουμε στο ζήτημα. Για τη Βοσνία. Πολλοί από εσά τονίσατε δικαίως ότι πρόκειται για, μια, για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι αυτό που αποφασίστηκε σήμερα ήταν ότι το έγγραφο της ε, Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας ε, αποτέλεσε θετική συμβολή στη συζήτηση, αλλά υπήρχαν και συμβολές ε, από άλλες χώρες και η Κροατία πριν από ε, κάποιους μήνες είχε υποβάλει κάποιες προτάσεις, οι χώρες Μπενελούξ το ίδιο, οπότε ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να συντονιστούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε. Αλλά πάντως ε, υπήρξε σήμερα μια κοινή αντίληψη από τα κράτη-μέλη με βάση την οποία φαίνεται ότι θα πρέπει να ξαναναλάβουμε την πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο ζήτημα, να μην το αφήσουμε επίσης μας. Και δεύτερον υπάρχει ε, μία... Ε, ε, ότι ενδεχομένως ο σωστός δρόμος είναι να δημιουργηθούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για το Παλαιστινιακό ζήτημα, αυτό που είπε η ύπατη εκπρόσωπος, εκπρόσωπος περιγράφοντας την επίσκεψή της εκεί είναι πολλά. Η κατάσταση στη Γάζα εξακολουθεί να είναι δραματική παρά τις διευθυντήσεις και τους διακανονισμούς που έχουν γίνει μεταξύ των Ισραηλινών αρχών και των αρχών του ΟΗΕ η ανοικοδόμηση της Γάζας προχωρά πάρα πολύ αργά και ένας από τους λόγους ε, ε, είναι ότι ο διακανονισμός εφαρμόζεται πολύ αργά. Αλλά επίσης ε, ένας από τους λόγους για την κατάπαυση των εχθροπραξιών ε, στη Γάζα ήταν για να μπορέσει η Παλαιστινιακή Αρχή να επανέλθει ως αρχή, ως εξουσία στην Γάζα. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί ε, ε, ε, εξακολουθεί να υπάρχει διαχασμός μεταξύ της Παλαιστινικής Αρχής και της Χαμάς. Και αυτός είναι ο λόγος που προς το παρόν δεν μπορούμε να, πούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχία. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πούμε και να κάνουμε ως συμβολή είναι να συνεχίσουμε να συζητούμε με τους εταίρους μας βεβαίως, με τους Αμερικανούς, γιατί ο Τζον Κέρι όπως γνωρίζετε αναλογίζεται ίσως το ενδεχόμενο να ξανανοίξει μια νέα πρωτοβουλία με την τετραμερή που συναντάται που προσπαθεί να δει αν μπορεί να αναλυθεί πρωτοβουλία από την τετραμερή, συζητεί με Άραβες της περιοχής για να δει αν μπορούν οι αραβικές χώρες να αναλάβουν μια νέα πρωτοβουλία όπως αυτή του σχεδίου της Βηρητού του 2002 που έχει πέρασει αρκετό καιρός μένα, αλλά επανέρχεται και θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή βάση για να συνεχίσουν από εκεί οι συνομιλίες. Αυτά λοιπόν και νομίζω ότι βλέπουμε εμείς από πλευρά μας, κοιτάμε πού μπορούμε να είμαστε πιο χρήσιμοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε ε, ένας παράγων που θα βοηθήσει, αλλά βέβαια όχι πιο σημαντικός. Ε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποτρέψουμε ένταση της βίας και περισσότερες, ε, περισσότερα προβλήματα. Η αναγνώριση τώρα. Η αναγνώριση είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Και εδώ θα πρέπει να γίνει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση μεταξύ της πρωτοβουλίας κάποιων ανθρικών κοινοβουλίων η οποία μπορεί να είναι διαφορετική από μια απόφαση της ίδιας κυβέρνησης για τη δική μου ας πούμε, χώρα που γνωρίζω καλύτερα. Ξέρουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες η Εθνοσυνέλευση θα συζητήσει, θα την ακολουθήσει το το, η Γερουσία, με αποφάσεις που ενδεχομένως θα ληφθούν, αλλά δεν θα σημάνουν απαραίτητα και αντίστοιχη κίνηση της κυβέρνησης. Αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες. Πάντως αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα η αναγνώριση όταν οι βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια δηλώνουν με την αναγνώριση μια τέτοια πρόθεση. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε σε αυτό γιατί δεν έχουμε και αρμοδιότητα. Πάντως, ή μη τι άλλο, θα κάνουμε όσο μπορούμε, ό,τι καλύτερο. Και έχουμε τις επαφές μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε. Λιβύη. Μια από τις τελευταίες ερωτήσεις. Με την κυρία Γκόμες. Για το αν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα τα κράτη-μέλη. Ναι, εγώ θα σας πω, ναι, την αντιλαμβάνονται, το πιστεύω πραγματικά και ανησυχούν ειλικρινά για τα συμβαίνονται εκεί. Η Μπερναρντίνο Λεουάνε, παραδείγματα, έχει οριστεί εκεί. μεταβαίνει, προσπαθεί να καταγράψει, να διατυπώσει διάφορες ιδέες. Λόγω όμως της έκτασης της βίας που εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή στη Λιβύη, θα πρέπει και να γνωρίσουμε ότι δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε στις συνθήκες τη δική μας παρουσία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στον έλεγχο των συνόρων λίγο πολύ, αλλά τα όσα συμβαίνουν στην Τρίπολη, την Βενγάζη, δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν διατηρήσει πρεσβείες, πρέπει να πω, στην Τρίπολη. Μάλιστα ένας από τους πρέσβες μόλις ενημερώθηκε από τις αρχές της Τρίπολης ότι πρέπει να αποχωρήσει. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, όλων μας, ότι τα συμφέροντα όλων μας μάλλον διακυβεύονται και πρέπει να σταματήσουμε. Στο σημείο αυτό οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι θα πρέπει να σταματήσουν λόγω υπέρβασης του ωραρίου. Ευχαριστούμε.